Right, good morning everybody. I think we have got every... Καλή σας μέρα. Νομίζω ότι τώρα εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές ομάδες. Ο για μαφίγει ο Πίτερ, άμα φύγει ο Πίτερ δεν... Α. If we can start, we uh, are on to θα ήθελα να αρχίσουμε το σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τωμάζο Παντόα Σκιώπα, που είναι πρόεδρος του Ιδρύματος Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ο οποίος ε, διαδέχθηκε τον προηγούμενο πρόεδρο στη... τον Ιούνιο, τον περασμένο Ιούνιο Ξέρετε ότι ο κύριος Παντοασκιώπα ήταν ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέχρι το 2005 και το 97-98 ήταν πρόεδρος της Κόνσορ έχει ε, επίσης διατελέσει σε πάρα πολύ γνωστές άλλες θέσεις υποθέτω ότι τον γνωρίζετε όλοι δεν χρειάζονται άλλες εισαγωγές και του δίνω αμέσως το λόγο για να έχουμε χρόνο για ερωταπαντήσεις Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε σήμερα εδώ. The ότι το θέμα ήταν τόσο ε, ενδιαφέρον που θα ήταν γεμάτη η αίθουσα σήμερα το πρωί. Δεν συμβαίνει αυτό βέβαια, αλλά θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κάνω μια σύντομη αλλά ενδιαφέρουσα παρουσίαση για αυτούς που κατάφεραν να έρθουν. Η δημιουργία διεθνών λογιστικών προτύπων είναι ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια που έχουν ποτέ αναλυφθεί στον τομέα της δημιουργίας κανόνων για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά άλλα αντίστοιχα projects είναι η απελευθέρωση του τραπεζικού τομέα, ε, διευθέτηση των τίτλων, ε, πολλοί, πολλοί τομείς ακόμη στους οποίους ε, διεθνείς επιτροπές στο παρελθόν προσπάθησαν να εφεύρουν, να αναπτύξουν κοινούς κανόνες. Τώρα τα λογιστικά δεν είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ενδεχομένως αλλά είναι ο νεότερος τομέας και ο πιο επιτυχημένος θα έλεγα το Ίδρυμα του οποίου προεδρεύω δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια όταν α, η Επιτροπή Βασιλείας άρχισε να λειτουργεί πριν από 35 χρόνια και άλλα ιδρύματα επίσης παλιά. Παρόλο όμως που το ίδρυμα αυτό της Επιτροπής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι νεαρό σε ηλικία έχει επιτύχει πάρα πολλά πράγματα στη σύντομη ζωή του. Σήμερα Υπάρχει ένα ολόκληρο σύνολο λογιστικών κανόνων που εφαρμόζονται άμεσα και που τηρούνται από πάνω από 180 χώρες. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σε κανένα άλλο τομέα. Ο λόγος για αυτήν την εντυπωσιακή επιτυχία είναι, οι λόγοι είναι πολλαπλοί. Πρώτον, το ίδρυμα που φτιάχνει αυτά τα λογιστικά πρότυπα που παλιά ονομαζόταν η Ask Foundation έχει ένα θεσμικό προφίλ το οποίο το καθιστά πιο αποτελεσματικό από άλλες επιτροπές σε άλλους τομείς στο τραπεζικό τομέα, στους κανόνες για το, για το τραπεζικό σύστημα κτλ. Το... Είμαστε ένα μικρό σώμα 15 ατόμων που δουλεύουμε με πλήρη ανεξαρτησία. Δεν είμαστε μέλη ενός συμβουλίου. Ο που προσπα, όπου προσπαθεί ο καθένα να υποστηρίξει τα εθνικά πρότυπα ε, και να προχωρήσει σε εναρμόνιση των ε, διαφόρων συστημάτων, όχι. Είμαστε πλήρως αφιερωμένοι στην ανάπτυξη διεθνών λογιστικών προτύπων εξ Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άλλος παράγοντας που οδηγεί σε επιτυχία είναι ότι το 2002 όταν το Ίδρυμα ήταν ακόμη στα Σπάργανα ε, η Κομισιόν έκανε μια την πρόταση να δημιουργήσει ένα ειδικό σώμα για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ε, και το, το θέμα πήγε στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και έτσι ε, ε, φτιάχτηκε, αναλάβαμε να φτιάξουμε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα τα οποία είναι υποχρεωτικά για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση για υποχρεωτικά λογιστικά πρότυπα του άμεσα εφαρμόσιμα ε, το 2002 επέλυσε ένα διέξοδο που πολλών δεκαετιών που κολυσιεργούσε αν θέλετε και αναχέτιζε ε, πολλές ε, διαδικασίες ε, και πολλές εγκρίσεις είχαν φτιαχτεί βέβαια κάποιες ε, ε, είχαν εγκριθεί κάποιες οδηγίες και τα λοιπά αλλά τα πράγματα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν τρίτος παράγοντας επιτυχίες ήταν το εξής ότι κάποιες αναδιόμενες οικονομίες οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο θεώρησαν ότι θα ήταν ε, καλό να εγκρίνουν άμεσα διεθνή λογιστικά πρότυπα αντί να ε, προσκοληθούν αν θέλετε σε στα αμερικανικά πρότυπα ή σε άλλα πρότυπα. Αυτή ήταν η κατάσταση στην οποία βρήκα το Ίδρυμα Διεθνών ε, Λογιστικών Προτύπων όταν άρχισα να δουλεύω τον περασμένο Ιούλιο. Το 2005 και 2006 είχα εργαστεί για το Ίδρυμα αλλά μετά όταν έγινα μέλος της τελικής κυβέρνησης εγκατέλειψε εκείνη τη θέση. Ανέλαβα λοιπόν τον Ιούλιο, βρήκα και βρήκα το Ίδρυμα μετά από 10 χρόνια να έχει επιτύχει πολλά. Αρχίζει όμως τώρα η δεύτερη δεκαετία ζωής του Ιδρύματος και ο αριθμός των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε για τα, τους επόμενους 12-24 μήνες είναι πάρα πολλές. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των προκλήσεων. Η θα επιτύχουμε πλήρη εντοποίηση και θα έχουμε παγκοσμίω ένα σετ λογιστικών προτύπων ή θα αναγκαστούμε να πισωγυρίσουμε και να εγκαταλείψουμε τις επιτυχίες της πρώτης δεκαετίας πράγμα το οποίο δεν είναι εναλλακτική λύση λοιπόν έγκριση των προτύπων ε, ποιότητα των ε, προτύπων και διακυβέρνηση του θεσμού αυτή είναι η τρεις βασική μας στόχη. έγκριση, adoption, υιοθέτηση των προτύπων τι εννοούμε εννοούμε όχι απλώς εναρμόνιση των εθνικών προτύπων, αλλά εξυπαρχής ε, υιοθέτηση νέων διεθνών προτύπων. Η στις Ηνωμένε Πολιτείε. Παραδείγματο χάρη του χρόνου πρέπει αυτέ να αποφασίσουν κατά πόσον από το ο, GAP να προχωρήσουν από το GAP στο FRS και η σχετική επιτροπή θα αποφασίσει το δεύτερο εξάμεινο μάλλον του 2011 για τα την έγκριση του ΑΕΦΑΡΕΣ ε, αυτό δεν σημαίνει άμεση θέση σε ισχύ των νέων προτύπων, αλλά θα ξέρουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2011 αν οι Ηνωμένε Πολιτείες θα πουνε ναι ή όχι. Αν πουνε ναι, περιμένουμε και προσδοκούμε ότι οι, την Ηνωμένε ε, Πολιτείε θα ακολουθήσουν και η Ιαπωνία και άλλες χώρες. Τώρα, το δεύτερη πρόκληση, ο δεύτερος στόχος είναι η ποιότητα. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ποιότητα των προτύπων αντικατοπτρίζει πλήρως τα μαθήματα τα οποία εξάγονται από την οικονομική κρίση, την σοβαρή οικονομική κρίση που μερικοί την συνδέουν και με κάποιες πτυχές των προτύπων και θα πρέπει να φροντίσουμε ότι είναι διεθνείς όχι μόνο οι κανόνες αλλά και οι εφαρμογή τους, ότι είναι συνεπής ομοιόμορφη η εφαρμογή τους, ώστε να μην υπάρχει ε, διολίσθηση, απόκληση κάποιων στην εφαρμογή. Τρίτος στόχος και πρόκληση είναι η διακυβέρνηση. Το ίδρυμα που δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια με βάση αμερικανικό, το αμερικανικό μοντέλο ε, ιδιωτικής, ιδιωτικού οργανισμού με στόχο δημόσιο συμφέρον και το οποίο διοικείται από ένα συμβούλιο τραστής, board of trustees. Αυτό το ίδρυμα λοιπόν που βασίστηκε σε αυτό το μοντέλο όταν ιδρύθηκε δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό. Ε, συνεχώς ζητείται η καλύτερη, η μεγαλύτερη νομιμοποίηση αν θέλετε αυτού του Ιδρύματος έγιναν πολλές μεταρρυθμίσεις για να αυξηθεί και η νομιμότητα και η λογοδοσία του Ιδρύματος αλλά με ένα τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να μην υπονομευθεί η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του Ιδρύματος βεβαίως το θέμα αυτό ακόμη εκρεμεί ε, βεβαίως εκτός από τον Board of Trustees υπάρχει και ένα εποπτικό σώμα, Monitoring Board, στο οποίο συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά βεβαίως όλα... Ε, για αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται δύο αναθεωρήσεις της στρατηγικής του Ιδρύματος από το Board of Trustees και από το Monitoring Board δύο αναθεωρήσεις λοιπόν οι οποίες βεβαίως για ε, αυτή τη στιγμή καταρτίζονται με στενό συντονισμό και συνεργασία. Ε, εν ώψη αυτών των αναθεωρήσεων λοιπόν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να πάρθει και μια απόφαση για τη μελλοντική διοίκηση και διακυβέρνηση του Ιδρύματος. Το Board of Trustees ετοιμάζει μια αναθεώρηση που αναφέρεται στην ποιότητα και στην ποιότητα των προτύπων και στην χρηματοδότηση του Ιδρύματος. Να πω δύο λόγια κλείνοντας για τη χρηματοδότηση γιατί αυτό είναι σημαντικό και αφορά και σας Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος αυτή τη στιγμή εν μέρη προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζουμε να εγκρίνεται την ε, συνεισφορά στη χρηματοδότηση του Ιδρύματος IFRS αλλά αυτή δεν είναι η μόνη χρηματοδότηση από την Ευρώπη η εθνική χρηματοδότηση στα θα συνεχίζεται στο βαθμό που θα υπάρχει κενό αν θέλετε μεταξύ των ποσών που δίνονται από το προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συνολικού ποσού που θα έπρεπε να προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει κλίδας που ορίζει τη χρηματοδότηση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή από την οποία αυτή προέρχεται. Θα ήθελα να κλείσω εδώ για να έχουμε χρόνο για έρωτα απαντήσεις. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολλής. Τις ομιλητές έχω λοιπόν στον κατάλογο. Δεν ξέρω αν θέλει και κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. So, Sven, list anyway. Ο Σβέν είναι ο πρώτος στον κατάλογο. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ και ζητώ συγγνώμη. Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε καλύτερα, να έχουμε δηλαδή μεγαλύτερη παρουσία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσέλευσή σας. Εγώ έχω μία σειρά ερωτήσεων. Στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για τους κανόνες που διέπουν την Επιτροπή ε, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων έχουμε θίξει δύο ζητήματα που θα πρέπει να εισαχθούν το συντομότερο δυνατόν στα πρότυπα αυτά. Θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορείτε να ε, εξασφαλίσετε, εξασφαλίσετε έτσι ώστε το Κοινοβούλιο συμμετάσχει στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων του σώματός σας και δεύτερον πώς θα ανταποκριθείτε στις επαναλημμένες εκκλήσεις και αποφάσεις αυτού του σώματος για να κινηθείτε ε, χώρα προς χώρα στην εφαρμογή κανόνων. Ιδιαίτερα στο τομέα των ε, κατασκευών, των βιομηχανιών και πώς θα ισχύσει η έκθεση χώρα προς χώρα. Γιατί θέλουμε τα λογιστικά πρότυπα να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Και εσείς ε, θίξατε θέματα νομιμότητας στη διάρθρωση του Ιδρύματος. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα δούμε πώς θα ανταποκριθείτε σε αυτό το αίτημα που προέρχεται από τις κυβερνήσεις αλλά και από μη κυβερνητικές. Ευχαριστώ. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για τις ε, δύο αυτές ερωτήσεις. Θα τις απαντήσω και τις ε, δύο και θα ζητήσω από το ε, συνεργάτη μου συμπληρώσει το δεύτερό σας ερώτημα, την απάντηση δηλαδή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, ελέγχει και ποπτεύει την εργασία του Ιδρύματος. Εμείς προβαίνουμε σε διαβουλεύσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με αυτό το σώμα, αν μας το ζητήσετε. Και έχουμε, λαμβάνουμε πολλά στοιχεία σε σχέση με τους διαχειριστές και το Ίδρυμα καθεαυτό ως προς το, ε, την Συμβουλευτική Επιτροπή. Όταν μιλάτε για λήψη αποφάσεων υπάρχουν πολλά επίπεδα λήψης αποφάσεων. Τα ίδια τα πρότυπα ορίζονται ε, από το ISB αυτόνομα. Οι διαχειριστές δεν ορίζουν τα πρότυπα αυτά Υπάρχει ειδικό input, μπορεί να γίνουν συστάσεις, υποδείξεις, αλλά όπως είπα και στην αρχική μου ε, παρουσίαση, το Συμβούλιο είναι ένα ανεξάρτητο σώμα και εκεί έγκυται και η επιτυχία του. Σημαίνει δηλαδή ότι κανένας δεν μπορεί να του υποδείξει τι να κάνει. Αυτά όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως και το Κογκρέσο της ΗΠΑ αντίστοιχα εκφράζει απόψεις και προβαίνει σε συστάσεις, αυτό εντάσσεται στην όλη διαδικασία και είναι μια πολύ καλή και ευπρόσδεκτη πρακτική. Ως προς τις εκθέσεις αναχώρα γνωρίζω αυτό το θέμα, τη σημασία του και έχει μεγάλη σημασία η δημιουργία προτύπων, διότι μιλάμε για διεθνή συνεργασία και βεβαίως και οι επενδυτές προβαίνουν σε επενδύσεις Τώρα, η κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανησυχίες, πολύ σημαντικές, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν παρέχουμε πληροφορίες τους ε, ενδυνάμει επενδυτές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς ορίζονται τα έσοδα και ποιος είναι ο συσχετισμός βιομηχανιών σε σχέση με τις ε, κεντρικές κυβερνήσεις και τη συνεργασία του βιομηχανικού τομέα. Βεβαίως μπορεί να γίνει διαφορετικός επιμερισμός αναχώρα και αυτό που προσπαθούμε είναι να ε, διατυπώσουμε ένα παρόμοιο αίτημα με αυτό που εντάσσεται στην Αμερικανική νομοθεσία μέσω του νομοθετήματος Ντόντα Φρανκ και ο συνάδελφος μπορεί να προσθέσει ορισμένα στοιχεία. Ευχαριστώ. Υπάρχουν τρεις τάσεις ως προς την ε, κατάσταση της κάθε χώρας καταρχήν ο κανόνας, μάλλον η διαχείριση των εξορρυκτικών βιομηχανιών. Εδώ υπάρχει ένα ειδικό έγγραφο, ένα ειδικό κεφάλαιο που αφορά το «Publish what you pay» ως προς τις εξορρυκτικές δραστηριότητες και βιομηχανίες. Είχαμε μία σειρά απαντήσεων μετά από ε, συναντήσεις με τους ε, εμπλεκόμενους φορείς και τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει αυτές τις επιστολές για να δει πώς θα διαχειριστεί το θέμα. Αυτό ως προς τις ε, εξορρυκτικές δραστηριότητες. Ο, ως προς το ίδιο το Ίδρυμα ορίζουμε τα διάφορα χρηματοδοτικά δελτία χρηματοπιστωτικά δελτία και όπως είπε και ο Πρόεδρος, αυτή τη στιγμή γίνεται μία αναθεώρηση στρατηγικής και στόχος του ε, Ιδρύματος είναι να ξαναδούμε τις προτεραιότητές μας ως προς τις υποδείξεις αναχώρα. Αυτό θα επηρεάσει αυτή την ε, αναθεώρηση. Η νομοθεσία τότε φρανκ ε, απαιτεί νέες αποκαλύψεις για τις εξορρυκτικές ε, δραστηριότητες μέσα στα πλαίσια ε, ενός μεγαλύτερου διάκαινου το οποίο θα πρέπει να καλυφθεί. Και νομίζω... Στα πλαίσια του GAP και αυτό που έχει σημασία είναι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να διαχειριστούμε το όλο πλαίσιο. Thank you, uh, Peter. Peter. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Άκουσα με ενδιαφέρον και το ίδιο και συνάδελφοι υποθέτω ότι η SEC θα προχωρήσει στη σύσταση του πλήρους IFRS. Έχουμε κάνει πολλές κοινοβουλευτικές αποστολές, έχουμε συναντηθεί με το Μέριο Σπύρο και άλλους ε, και ε, βλέπαμε τα αποτελέσματα του πρώτου, του δευτέρου εξαμήνου της τάδε χρονιάς για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και απογοητευτήκαμε γιατί την κρίσιμη ώρα δεν έκαναν αυτά που είχαν πει ότι θα κάνουν. Σήμερα φαίνεται ότι έχετε μεγαλύτερη πειθαρχία από αυτά που μας είπατε δηλαδή και εγώ δεν αισθάνομαι την ίδια αυτοπεποίθηση, πολύ θα χαρώ αν αληθεύει αυτό. Θα δούμε. Ε, και υπάρχουν και οι ενδιάμεσες εκλογές ε, και το νομοσχέδιο Dodd Frank που αναφέρατε ε, φέρνει αυτό ριζικές αλλαγές στη ΣΥΠΑ, οπότε ενδέχεται να απορριφθούν οποιαδήποτε δαπά πρότυπα, ας τα πούμε έτσι. Today, ε, Σήμερα ε, το IFRS είναι τα πλέον αποδεκτά διεθνή πρότυπα, δηλαδή ανά τον κόσμο, ε, και η Ευρώπη τα χρησιμοποιεί, αλλά όχι μόνο, και η Ασία. Αν δείτε τώρα την ε, συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς ε, για τις καταχωρημένες στο χρηματιστήριο εταιρείε. που οφείλουν να εφαρμόζουν συγκεκριμένα λογιστικά πρότυπα, το μερίδιο των ΙΠΑ φθήνει. από τα δύο τρίτα έχει φτάσει στο ίμιση περίπου στη, ως προς την παγκόσμια δηλαδή κεφαλαιοποίηση της αγοράς λόγω ε, των νέων μεγάλων ασιατικών εταιριών που χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα IFRS. Οπότε ε, τα, δεν είναι πλέον τα αμερικανικά πρότυπα, τα παγκόσμια πρότυπα δεν, δεν είναι πλέον σε θέση ισχύω ούτως ώστε να αναδειχθούν σε πρότυπα αναφοράς για τις εταιρείε. Οπότε για τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείε ε, είναι επιτακτική ανάγκη να ε, προσχωρήσουν στο IFRS ε, και θα δημιουργήσουν έτσι μια κρίσιμη μάζα ούτως ώστε να εγκριθούν αυτά τα πρότυπα. Ε, νομίζω ότι η απόφαση θα είναι θετική ε, λόγω αυτού και βασίζω την πεποίθησή μου σε επανειλημμένες επαφές που είχα το τελευταίο εξάμεινο, τα τελευταία, ε, τους τελευταίους πέντε μήνες στο Συμβούλιο των Διαχειριστών του Καταπιστεύματος με τις Αμερικάνικες Αρχές και τον πρόεδρο του ISCC και το IFRS. δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη την απόφαση. Η ISCC σαφέστατα τάσεται υπέρ, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το περιβάλλον που ισχύει στη ΣΥΠΑ, ε, στο Κογκρέσο, στον επιχειρηματικό κόσμο ή στην Αμερική γενικότερα. Ε, αληθεύει ότι αν οι ε, παρότι οι μεγάλες εταιρείες είναι σαφώς υπέρ ή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν μικρότερο διεθνή προσανατολισμό τείνουν να μην συμφωνούν όπως οι μεγάλες εταιρείες. Η φυστάμενη δομή για τα πρότυπα, τα FASB δηλαδή και το FIF, e το Ίδρυμα δηλαδή, ε, που είναι το αντίστοιχο του Ιδρύματος IFRS, ε, αναρωτιούνται ποιος θα ήταν ο ρόλος τους εάν τελικά ε, εγκρίνονταν τα πρότυπα του IFRS και πάλι είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους επανειλημμένα ε, συναντήθηκα με τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του IFRF, του Συμβουλίου Διαχειριστών του FIF, συγγνώμη, Οπότε θα είναι δύσκολο να ληφθεί η απόφαση στη ΣΥΠΑ. Κατά πάσα πιθανότητα σας λέω θα είναι θετική η έκβαση, αλλά η εφαρμογή θα είναι σταδιακή. Συν το χρόνο θα γίνουν και οι προσαρμογές που χρειάζονται. Κατά πάσα πιθανότητα ε, θα αρχίσουν με το να καταστήσουν εφαρμοστέα τα πρότυπα το AFRS ε, για τις μεγάλες εταιρείες σε πρώτη φάση. Εγώ ε, θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο πιθανή έκβαση, αλλά δεν αποκλείω και μια αρνητική ε, έκβαση και έχω πλήρη επίγνωση του ότι ε, αν τελικά είναι αρνητική η απόφαση, αυτό επισύρει μια σειρά συνεπειών για το IFRS η διακυβέρνησή του, η σύνθεση των οργάνων του, παραδείγματος χάρη και ο τρόπος λειτουργίας του Ιδρύματος, γιατί η ISB έχει δομηθεί ως ένα διεθνές ε, πρότυπο, εκπόνηση, ε, ε, κέντρο εκπόνησης προτύπων, ενώ ο, ο κόσμος όλος δεν ακολουθεί απαραίτητα το IFRS και με κάποιο τρόπο πρέπει να καλύψουμε το, το κενό και ελπίζουμε ότι με την ευρύτερη αποδοχή και έγκριση των προτύπων θα καλυφθεί αυτό το κενό. Υπερβάως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απάντησή σας προς το Σβέν Γκίγκολ καταδεικνύει την ε, δυσκολία που αντιμετωπίζουμε για αυτά τα λαγιστικά πρότυπα ως προς την εκπόνησή τους δηλαδή και το ρόλο τους στη διακυβέρνηση μας. Είπατε ότι ε, το βασικό αντικείμενο του ASB είναι η εκπόνηση προτύπων που είναι χρήσιμα για τους επενδυτές. Όμως, Βλέπουμε ότι είναι πανταχού παρόντα αυτά τα πρότυπα στην, στο δημόσιο διάλογο, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά διεθνή πρότυπα. Αυτά είναι. Ε, οπότε έχουν καταλητική σημασία για όλους τους εταίρους, είτε το θέλουν είτε όχι. Ε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουμε το πρόβλημα με την υποβολή εκθέσεων αναχώρα. Ε, και εδώ μιλήσαμε για την εξωρεκτική βιομηχανία, για τις ενδιαφερόμενες χώρες, κυρίως τις πτωχότερες εξ αυτών, αλλά ε, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος προσέγγισης ε, των παγκοσμίων προκλήσεων, δηλαδή χρηματοπιστωτική σταθερότητα ε, και ο προκυκλικός χαρακτήρας, ενδεχόμενος προκυκλικός χαρακτήρας αυτών των προτύπων. Και συχνά αναρωτιούμαστε το εξής. Εάν ε, στα πλαίσια μιας ε, καλά οργανωμένης παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, που βέβαια ακολουθεί μια μεταρρύθμιση στον δρόμο που χάραξε η G20 και θα μας πείτε αν μπορούμε να έχουμε ελπίδες, δεν μπορούμε να φανταστούμε μια πιο στενή διασύνδεση όπως το είχαμε πει και στο Κοινοβούλιο ανάμεσα στο ISB το Ίδρυμά της δηλαδή και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι μία από τις ιδέες που διερευνήσαμε εμείς και ποια απάντηση δόθηκε ε, η σύσταση αυτού του Συμβουλίου Παρακολούθησης. Πλην όμως έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το Συμβούλιο Παρακολούθησης εποπτείας δεν μας επιτρέπει να βγούμε από αυτή τη λογιστική λογική που παρόλα αυτά έχει επιπτώσεις που υπερβαίνουν τις ίδιες ανησυχίες των ε, λογιστών. Δεύτερη ερώτηση. Τι πιστεύετε για την εκπροσώπηση των Ευρωπαίων στα πλαίσια όλου αυτού του μηχανισμού. Δηλαδή, μόνο και μόνο το ότι ε, υπάρχουν κάποιες συμμετοχές στην ομάδα εποπτείας ε, επαρκεί και έχω και άλλες δύο ανησυχίες που θα ήθελα να εκφράσω. Πρώτον, η διαδικασία διορισμού. Είτε μιλάμε για τους διαχειριστές του Συμβουλίου, του καταπιστεύματος και θεωρείτε ότι η διαφάνεια, η νομιμοποίηση είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα. Ε, και δεύτερον, πάλι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ε, για την, ε, το διάλογο περί εύλογης αξίας, συνεχίζεται ο διάλογος ε, για την ευλογία αξία ε, και ε, επίσης για τα νέα πρότυπα που συζητούμε τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυρίως μετά τις εργασίες της, του Συμβουλίου της Βασιλείας είναι βέλθα τα αποτελέσματα σε σχέση με τους στόχους μας, αναρωτιόμαστε. Μπορούμε ταυτόχρονα να κατοχυρώσουμε το ότι θα είναι βανάγνωστοι οι λογαριασμοί, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουμε και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα βελτιστοποιούμε και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ε, Merci, euh, Madame Beres, pour Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις ε, ερωτήσεις. Τέσσερις πολύ σημαντικές ε, ερωτήσεις. Θα αρχίσω από την τελευταία και θα καταλήξω με την πρώτη. Είναι γεγονός ότι τα πρότυπα έχουν επινοηθεί καταρχήν για να εξασφαλίσουν ε, την πληροφόρηση των επενδυτών. Έτσι έχουν ε, επινοηθεί. Το, το ίδιο ισχύει για το US GAP, για το IFRS και ούτω καθεξής. Αφορά όλα τα πρότυπα ανά τον κόσμο. Υπάρχει ε, δημόσιο ενδιαφέρον, δηλαδή οι επενδυτές θα πρέπει να πληροφορούνται, αλλά υπάρχει και δημόσιο ενδιαφέρον για την ε, οικονομική σταθερότητα και για την γενικότερη υποστήριξη ως προς τους φυσικούς πόρους και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό θέλουμε να εξασφαλίσουμε και για κάθε στόχο ίσως ε, τα, τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης να μην είναι τα ίδια με μία άλλη. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε λογιστικά πρότυπα για την πληροφόρηση των επενδυτών που να είναι διεθνή, καθαρά διεθνή, που να μην αφορούν ε, συγκεκριμένους τομείς και να ισχύουν ε, για όλους τους ε, τομείς ή τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις και πρέπει να είναι ουδέτερα σε σχέση με τα επιχειρηματικά πρότυπα ενό συγκεκριμένου τομέα. Δηλαδή στον τραπεζικό τομέα υπάρχουν διάφορα business models και μερικά καταδεικνύουν ότι αυτά τα πρότυπα ευεργετούν συγκεκριμένους τομείς σε σχέση με άλλους. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχουμε λογιστικά πρότυπα τα οποία να έχουν μία ε, ιδεώδη, ας το πούμε, ιδεατή ε, κατάρτιση που να προβάλλουν κάτι άλλο πέρα από την πληροφόρηση του επενδυτή, δηλαδή προστασία φυσικών ε, πόρων, ε, προστασία της βιομηχανίας και ούτω καθεξής. Όταν βρισκόμουν στον τομέα των ρυθμίσεων και ρυθμιστών, τότε ε, μου έλεγαν ότι οι ρυθμιστές ορίζουν τα δικά τους ε, πρότυπα που ισχύουν για την ε, πληροφόρηση των επενδυτών. Οι επόπτες, οι εποπτικές αρχές δεν ήταν αυτή της άποψης οι δικοί μου συνάδελφοι. Για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι ότι έχουν πια προσλάβει τέτοια σημασία οι χρηματοπιστωτικές αγορές που κανένας δεν τολμά να διατυπώσει πρότυπα που να βασίζονται από, σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά της αγοράς. Κατά την άποψή μου αυτό είναι λάθος, αλλά πρόκειται για ένα λάθος το οποίο δεν ε, την χάνει αναγνώρισης, έτσι ώστε να διαφοροποιήσουμε τα πρότυπα. Άρα, οι επόπτες και οι θεματοφύλακες της οικονομικής σταθερότητας προσπαθούν να πείσουν τους standard setters, όπως το ISB, να λάβουν υπόψη αυτή τη διαφοροποίηση. Και τα τελευταία πρότυπα του ISB για τον χρηματοοικονομικό κόσμο λαμβάνουν υπόψη την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα χωρίς να υπάρχει ε, ανέλικτη ερμηνεία του fair value και προσπαθούμε να προσανατολιστούμε αλλού και αλλού. Δηλαδή να φτάσουμε σε μια εξισορρόπηση όλων των συνιστοσών. Και αυτό ακριβώς γίνεται. Όσον αφορά την ε, διαφάνεια, ο πιο πρόσφατος διορισμός αφορά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός έγινε μετά από ενδελεχή ε, έρευνα των υποψηφιωτήτων και μετά από διαβούλευση του Monitoring Board που δεν προβλεπόταν αρχικά αλλά έγινε και συνεισέφερε στο τελικό αποτέλεσμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό όχι μόνο για τους διαχειριστές καταπιστεύματος αλλά και για το Monitoring Board, το ελεγκτικό συμβούλιο, εποπτικό συμβούλιο. Εάν πρέπει να συγκρίνω το διορισμό, με τους διορισμούς σε άλλα σώματα όπως η ΕΚΤ δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει επαρκής λογοδοσία στο δικό μας Ίδρυμα και διαφάνεια. Νομίζω ότι το Συμβούλιο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, το Financial Stability Board, αυτό ακριβώς προβλέπει. Και θέλουμε να δώσουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα στον κόσμο ως προς την εκπροσώπηση των Ευρωπαίων στο Ίδρυμα αυτόν. Επαναλαμβάνω, έχουμε να κάνουμε με μία ε, αρχιτεκτονική που αφορά την παγκόσμια εκπροσώπηση ανεξάρτητα από από την έγκριση των, προτύπων, των στη μία ή στην άλλη χώρα. Υπάρχει δηλαδή υψηλή παρουσία Αμερικανών στους διαχειριστές, αν και το IFRS δεν έχει εγκριθεί στις Ιπα. Μπορούμε να αντιταχθούμε βεβαίως σε κάτι τέτοιο. Και εάν υπήρχε αρνητική στάση γενικά των Ιπα, αυτό θα είχε συνέπειες εάν βρισκόμασταν στην αντίστροφη κατάσταση, δηλαδή το Standard Setting Body των ΙΠΑ ήταν το αντίστοιχο του, που εκπροσπούσε τον κόσμο και οι Ευρωπαίοι εκπροσωπούνταν αλλά δεν δέχονταν τον καθορισμό των προτύπων, θα λέγαμε ότι πρόκειται για ε, ένα δείγμα αμερικανικού ιμπεριαλισμού που δεν μπορούμε να δεχτούμε. Άρα αυτή η εκπροσώπηση, κατά την άποψή μου, δεν είναι λανθασμένη. Όμως η ευρωπαϊκή παρουσία μεταξύ των τραστής, των ε, διαχειριστών, στα πλαίσια του ε, συμβουλευτικού συμβουλίου δεν δείχνει ότι υπάρχει ε, έλλειψη παρουσίας Ευρωπαίων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πιστεύω ότι η διακυβέρνηση ε, διαρθρώνεται σε τρία-τέσσερα επίπεδα. Το ISB, τους διαχειριστές, το Monitoring Board και τους G20, οι οποίοι ασχολούνται με τις δραστηριότητες, τους στόχους και τα προγράμματα ως προς την κατάρτιση λογιστικών προτύπων. Το τρίτο επίπεδο, το Monitoring Board, απορρέει από το ΙΟΣΚΟ. Δηλαδή δεν του έχει αναθεθεί καμία εντολή από τους G20 που δεν, ήταν, ε, δεν είχαν λάβει δραστηριότητα εκείνη την εποχή και δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει νομιμότητα του Monitoring Board. Αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα που θα κρίνουμε εμείς. Θα το κρίνουν οι διαχειριστές καταπιστεύματος. Εν πάση περιπτώσει το Monitoring ε, Board ε, έχει τη δική του εργασία. Εγώ είχα διοριστεί με συνοπτικές διαδικασίες μία φορά στο Monitoring Board. Θα τελειώσω εδώ. Το Monitoring Board ε, τώρα αναθεωρεί τις βάσεις του, αναφέρεται στις, ε, στους διεθνείς οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάτι τέτοιο θα ήταν επιθυμητό αλλά δεν θα το αποφασίσουν οι διαχειριστές αλλά το Monitoring Board ή η G20 όπως και το IFRS είναι μια διεθνής οργάνωση για τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση τα ε, κλασικά όργανα τα οποία βασίζονται στις συνθήκες και έχουν πλήρη νομιμότητα. Κάτι τέτοιο αντίστοιχο ισχύει και για το Monitoring Board. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν και άλλοι δύο ομιλητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ όταν μιλήσαμε για το εποπτικό πακέτο και προσπαθήσαμε να εισαγάγουμε την αρχή του να ισχύουν λογιστικά πρότυπα αναχώρα, τότε είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ε, παγκόσμια λογιστικά πρότυπα, αλλά να βρούμε και επιπρόσθετες φόρμουλες που να σχετίζονται με πρότυπα σε, με βάση την κάθε χώρα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη που να απορρέουν δηλαδή από παγκόσμια πρότυπα για την χρηστή διακυβέρνηση. Γιατί τα πρότυπα μπορούν να συνεισφέρουν έτσι ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα και να φτάσουμε στους παγκόσμιους στόχους σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή, οι εταιρικές σχέσεις, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή, θα πρέπει να μην φτάσουμε σε μια χρηματοοικονομική ε, ανισορροπία και αν υπάρχουν ε, προβλήματα από πλευράς πιστωτών, τότε θα ανακύψουν ακόμα μεγαλύτερα θέματα ως προς την ε, ποιότητα. Θα ήθελα να πω τα εξής. Η ποιότητα βασίζεται σε ορισμένες αρχές ή προδιαγραφές. Καλύτερα να ε, βασιστούμε ίσως σε προδιαγραφές. Αυτό αφορά τον τομέα, τους επιμέρους τομείς. Όμως η αγορά χρειάζεται αρχές και όχι μία συνεταιριστική προσέγγιση. Αυτό θα επηρεάσει την χρηστή διακυβέρνηση, γιατί δεν θα πρέπει να είναι μία διακυβέρνηση ε, διαχειριστικού ή συνεταιριστικού χαρακτήρα, αλλά θα πρέπει να αφορά το σύνολο της αγοράς. Γι' αυτό τελικά οι τελικοί δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν διαφανείς πληροφορίες που να αφορούν τη διακυβέρνηση στο σύνολό της, μέσα στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών ή χρηματοπιστωτικών διεθνών ιδρυμάτων Πώς θα εξελιχθεί αυτή η πορεία κατά την άποψή σας. Ο Ιντάλγκο. Α, όχι, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ πολύ και σας, σας ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση που μας κάνατε. Ε, είμαι λογίστρια ε, και ασχολούμαι και με εσωτερικούς ελέγχους και προφανώς με ενδιαφέρουν αυτά τα ε, διεθνή πρότυπα. Ε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το 98% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μόνο 2% των επιχειρήσεων είναι μεγάλες. Η ε, εισαγωγή λοιπόν διεθνών προτύπων στη χώρα μου θα και σε άλλες χώρε, χώρες σε πάση περιπτώσει που εφαρμόζεται και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ήταν το κερασάκι στην τούρτα των ήδη πολύπλοκων λαφρεοκρατικών κανόνων που τους οποίους έπρεπε να τηρούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο βάρος για αυτές. Είναι τεράστιος ο φόρτος που καλούνται να αναλάβουν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι τα διεθνή πρότυπα ε, βοηθούν τις επιχειρήσεις αυτές. Από την οπτική γωνία λοιπόν της Ευρώπης και αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ενιαία εσωτερική αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη και σας λέω το μεγαλύτερο ποσοστό η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και τι τι όφελος έχουμε από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Πώς βοηθούμε με την εισαγωγή αυτών την εσωτερική αγορά. Τι μαθαίνουμε παραπάνω μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις των διαφόρων κλάδων αναχώρα, των διαφόρων χωρών μεταξύ τους ή όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση χρόνου. Γέμισε η αίθουσα από ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για τα λογιστικά πρότυπα αλλά είναι συντάκτες ε, θέσεων. Ε, σημείωσα τις, τα σχόλια του κυρίου Σαντζες, Ουσιαστικά η, ε, μίλησε για την προσέγγιση ε, αρχές υπέρ της, των αρχών και κατά των κανόνων. Των προτύπων βασίζονται σε αρχές και όχι αυτών βασίζονται σε κανόνες. Αυτή είναι μια φιλοσοφική, αν θέλετε, προσέγγιση ε, θεμητή η η ύπαρξη και των δύο προσεγγίσεων αλλά οι, αυτοί που εφαρμόζουν τα πρότυπα προτιμούν τους κανόνες από ό,τι φαίνεται είναι από πρακτικής απόψεως βολεύουν καλύτερα τα στάνταρ που βασίζονται σε κανόνες και ε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν δέχονται οι Αμερικανοί. Ε, τώρα, η κυρία Καλπέλς Μίλησε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Κοιτάξτε, υπάρχουν πρότυπα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, Επανειλημμένως έχω ζητήσει από το ISB όταν για πρώτη φορά έγινε πρόεδρος ε, του Board of Trustees πριν από πέντε χρόνια είχα ζητήσει επανειλημμένως να φτιαχτούν ειδικά πρότυπα για τις, SM, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που να είναι πιο απλά στην εφαρμογή τους. Δεν είναι βεβαίως υποχρεωτικά στην Ευρώπη ή, αλλά ε, εγώ θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία που χρησιμοποιείται ευρέω, αλλά δεν είναι υποχρεωτικά άρα δεν φορτί, δεν επιβαρύνουν δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να δώσω, σας δώσω μια ιδέα. Τα πρότυπα των, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από άποψη σελίδων είναι περίπου ένα δέκατο των σελίδων των κανονικών προτύπων. Κάναμε μια τεράστια, τεράστια προσπάθεια για να απλουστεύσουμε τα πράγματα και να είναι και πιο φτηνά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα τη σχέση μεταξύ των προτύπων και της ενιαίας αγοράς. Σημείο κλειδί για την ενιαία εσωτερική αγορά δεν είναι μοναχά η ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων αλλά και η οικονομική ενοποίηση με την αυρία έννοια αν θέλετε που ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει άμεσε άμεσες επενδύσεις ε, θα οδηγήσει σε περισσότερες κερδοφόρες επενδύσεις γενικότερα άσχετα από τα γεωγραφικά σύνορα ή τις διαχωριστικές γραμμές των διαφόρων οικονομικών κλάδων. Για να έχουμε ένα ενιαίο τρόπο να μετρήσουμε τις επιδόσεις κάποιας επιχείρησης και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το ενδεχόμενο επένδυσης σε κάποιο κλάδο ε, για κάποια επιχείρηση ε, μπορούμε κάλλιστα να χρησιμοποιήσουμε τα πρότυπα. Άρα υπάρχει πολύ στενή σχέση με την εσωτερική αγορά και την ε, την ε, ενιαία μέτρηση, ομοιόμορφα πρότυπα δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη για την ε, φασαρία που έγινε με τα ε, λόγω των ε, συναδέλφων που ήρθαν για να ψηφίσουν αλλά τουλάχιστον άκουσαν και μερικά πράγματα για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα έμαθαν και κάτι τι ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ κύριε Σκιώπα ε, και εγώ ευχαριστώ Right, everybody, we are going to be moving on to... Ας προχωρήσουμε λοιπόν στο σημείο 9 τώρα της σημερινής διάταξης. Ε, ψηφίζουμε για την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2009. Ελπίζω ότι φέρατε όλοι τις κάρτες σας αν υπάρχουν και μερικοί που έχουν πανικοβληθεί γιατί πήραν ότι, γιατί είδαν ότι δεν έχουν την κάρτα μαζί τους, να σηκώσουν το χέρι. Η Βίκη, μία. Πολύ καλά. Λοιπόν, αν οι ψηφοφορίε είναι... Α, ε, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Λοιπόν, ψηφίστε δοκιμαστικά παρακαλώ. We will find out which buttons you pressed. Yeah, Για να δούμε. We got okay. Plus is happy, 29. Only four minuses. Λοιπόν, υπέρ είναι <laughs> κατά 4 και διάφορες εποχές. Δουλεύει το σύστημα λοιπόν. Λοιπόν, Παράγραφος 1. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 2. Το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 1 καταπίπτει τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λύση γιατί ένα μέρος της είναι κίτρινο. Τέλος πάντων τροπολογία υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρα 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται okay. I'm amendment 21. Τροπολογία 21. Τελευταία στιγμή ζητήθηκε τη ψηφοφορία. Όχι, δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, τροπολογία 21, κανονική ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 ΙΜΚΟ εδώ ζητήθηκε χωριστή ψηφοφορία για τις λέξεις Opting Principle and Taking into Account the. Την έχετε αυτή την τροπολογία. Λοιπόν, ψηφίζουμε για το κείμενο πρώτα-πρώτα χωρίστε αυτές τις λέξεις και μετά ψηφίσουμε για τις λέξεις αυτές. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ του κειμένου δίχως τις λέξεις αυτές. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά έχουμε το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά, αποχές, Ωραία. Είμαστε υπέρ, είστε υπέρ κατά των λέξεων, ε? Το καταλάβατε τι ήθελα να πω. Ωραία λοιπόν. Λοιπόν, εγκρίνεται και το δεύτερο κομμάτι. Όχι, εγκρίνεται η τροπολογία δίχως τις λέξεις αυτές λοιπόν. We now a split vote on... Τροπολογία 22, χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος της 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πρώτο τμήμα, δεύτερο τμήμα λοιπόν υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα. Το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 22 για την οποία ζητήθηκε ψηφοφορία κατά τμήματα. I, I'm not voting, okay. okay. Right, that's carried. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβιβαστική πρόταση Β. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά καλύτερα να το επελευθεύσουμε 27 λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά Ψηφίσατε όλοι okay. That's carried. Εγκρίνεται λοιπόν Δίκιο είχα και πριν Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική λύση Γ Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 εμκό, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 παραγραφό του αρχικού κειμένου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εν, απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ούτως ή άλλως συμβαστική δέλτα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Amendment Τροπολογία 39 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Α, συγγνώμη. was adopted, η συμβαστική γάμα εγκρίθηκε όποτε αυτό καταπίπτει 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ. Κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε το 43 παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 47 καταπίπτει, 48 επίσης, 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. για την τροπολογία 50 μια αλλαγή της τελευταίας στιγμή. Προηγούμενα δεν είχαμε αποφασίσει αν θέλουμε developing ή evaluating. Τώρα η πρόταση είναι να πούμε developing and evaluating. Λοιπόν, η Σόφη το ζήτησε αυτό. Ε, ένα λεπτό. Ο κύριος Σάντσες Πρεσέντο το ζήτησε. Αλλά εντάξει, συμφωνώ. Λοιπόν, λοιπόν, με αυτή την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί 54 Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο λοιπόν της παραγράφου 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται και αυτή ε, το αρχικό κείμενο υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ το αρχικό κείμενο το original text της παραγράφου 14 Oh, right, so that's changed. Uh, that άλλαξαν τα πράγματα, εγκρίνεται. Βάση περιπτώσει. Τροπολογία 57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφης 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ εγκρίνεται 21 προς 20 το σκορ το αρχικό κείμενο της 17 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτό 62 καταπίπτει 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ήτρε 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές Επαλήθευση ηλεκτρονική παρακαλώ για την 88. Πέρες ψηφοφορία θα περίφθη τελικά. Η 88. Ποια ήταν αυτή η 88 αναρωτιέται η πρόεδρος. Τραν τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, μεταφορών 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, της Επιτροπής Μεταφορών 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 της Ιδίας Επιτροπής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η παράγραφος 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 της ΥΜΚΟ. υπέρ κατά. Για την ΥΜΚΟ 6 θα ήθελα να ξαναψηφίσουμε, δεν ξέρω τι κάνει το ΕΛΚ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 21, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπορούμε να επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα για την 65. 65. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. Το πρωτότυπο κείμενο για την παράγραφο 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 66 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται για την παράγραφο 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το πρωτότυπο της παραγράφου 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Α, Δεν ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Πάμε προς τα κάτω. Ήμκο 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 72 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η παράγραφος 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 73 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της 73. Ψηφίστε παρακαλώ. Okay, Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ήτρε 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα 26. Το δεύτερο τμήμα μόνο. Το δεύτερο τμήμα της 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήτρε 10. Υπέρ κατά. Τε, ξαναψηφίζουμε για την Ήτρα 10 υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά. Αποχές, επαλήθευση για την 74 παρακαλώ. vote, that's carried. Amendment 75 in... 75 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ο, η 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 16 υπέρ Έκανε λάθο η πρόεδρος, είναι ήτρε και όχι ΙΜΚΟ, 16 ήτρε υπέρ, κατά. Μπερδευτήκατε. Μπορούμε ομού να ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Όχι, ήτρε 16 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 18 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ήτρε 19 υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Το πρωτότυπο κείμενο της 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εντάξει επαλήθευση αν θέλετε για την 93 ψηφίστε παρακαλώ για την 93 κάνουμε την επαλήθευση Ψήφισαν όλοι, όντω εγκρίθηκε. Ήτρα 14 καταπίπτει και πάμε τώρα στην ΙΜΚΟ 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 13 με προφορική τροπολογία που προσθέτει το EG, λόγου χάρη δηλαδή, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τραν 18 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση παρακαλώ για την τραν 18. Εγκρίνεται. Τρέν 16 με προφορική τροπολογία αλλάζουμε το R advances και γίνεται benefiting from state support που από κρατική επιχορήγηση υπέρ παρα... κατά αποχές εγκρίνεται. ΤΡΑΝ 22 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται επαλήθεση για την Τρέν 22. Ψήφισαν όλοι. Όχι, εγκρίθηκε. Τραν 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τραν 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Την τραν 2, μια επαλήθευση σας παρακαλώ, τραν 2. Ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Βίκυ. Εκτός μικρόφων. Α, έχει την κάρτα της. Θα μπορούσε να είναι καταλητική η ψήφο όμως. Τέλος πάντων, απορρίπτεται γιατί είναι ισοψηφία 20 προς 20. Λοιπόν, επειδή υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 5 υπέρ κατά Αποχέ. Νομίζω ότι εγκρίνεται παλήθευση για την Τραν 5, παρακαλώ. Είναι σημαντικό να σηκώνετε το χέρι, ξέρετε, για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε. Ψήφισαν όλοι εγκρίνεται. Τραν 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 11 με προφορική τροπολογία το ascertain το κάνουμε assess και μετά διαγράφουμε το τελευταίο τμήμα της παραγράφου μαζί με την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τραν 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε ΙΜΚΟ 12 με προφορική τροπολογία το deregulation το κάνουμε opening. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίθηκε. Τραν 19 ε, υπέρ. Α, έχει καταπέσει. Τραν 20 υπέρ. Κατά. Δεν μου αρέσει να μετρώ μόνο το συντονιστές. Σηκώστε τα χέρια σας παρακαλώ. Τραν 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τράν 21, 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίση. Τράν 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ήτρε 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ήτρε 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ήτρε 23 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, ε, Τροπολογία 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το πρωτότυπο κείμενο 4 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Μπερδεύτηκα. Για την τροπολογία 9 παρακαλώ επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι οι απερίφθη. Το πρωτότυπο κείμενο το εκτιμώντας paper κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πρωτότυπο F, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πρωτότυπο G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το πρωτότυπο H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές αναφορές 1 15 πρωτότυπο κείμενο υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Ηλεκτρονικά η ψηφοφορία για το τροποποιηθέν κείμενο. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. 38 ψήφοι υπέρ και 2 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Επίνγκ. Κύριε Πίνκτη, θέλετε να πείτε κάτι. σα ευχαριστώ για την υποστήριξή σα. Θέλω να πω μόνο το εξή. Με αυτό το ψήφισμα ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει περίπου 15 μελέτε και ανασκοπήσει. Αν συμφωνείτε, θα παραμείνω σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε τι μπορεί να γίνει και πώ θα ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητέ μα και του σκιώδει θα του ενημερώνω διαρκώ για την πρόοδο που σημειώνεται. Ε, γιατί υπάρχουν πολλέ μελέτε που πρέπει να γίνουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ερευνητικό Ινστιτούτο, είναι όργανο εκπόνηση πολιτική. Σα ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο σημείο 10, δηλαδή ΑΕΠ και πέρα από αυτό η μέτρηση της πρόοδου σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο. Είσαστε έτοιμοι. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Χουντής, θέλει να μιλήσει παρακαλώ. Είστε το λόγο κύριε Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω απλώς να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους οι οποίοι δούλεψαν τις συμβιβαστικές λύσεις και τους ευχαριστώ για αυτή τη συμβολή και για αυτή την προσπάθεια και όπως φαίνεται από τη voting list με τις περισσότερες, αν όχι με όλες, συμφωνώ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ. Προχωρούμε στην ψηφοφορία. Συμβασμό α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμό Σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός Δ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Μπορούμε να ελέγξουμε όμως την 22. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πράγματι εγκρίθηκε. 23-24 καταπίπτουν. 25 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Μπορούμε να ελέγξουμε την 25 παρακαλώ. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Ισοψηφία. Άρα καταπίπτει. Απορρίπτεται μάλλον. Right. 26 um, σε δύο τμήματα με μία προφορική. Η προφορική είναι και στα δύο τμήματα. Τμήμα 1 υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας ελέγξουμε. Ελέγχουμε το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. I haven't because I'm not voting because they're all out there. Εγώ δεν ψηφίζω, λέει η πρόεδρος. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Καταπίπτει 27, 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός ε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 με προφορική υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 34. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πράγματι εγκρίνεται. Συμβασμός F υπέρ. F υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός G υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται ο συμβιβασμός G. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές. Μπορούμε να ελέγξουμε παρακαλώ την 43. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Συμβασμός H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47. Όχι, με συγχωρείτε, αι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτός ο συμβιβασμός, πρόταση συμβιβασμού. 48 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 49 έχει καταπέσει, 50 υπέρ, κατά αποχές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 με, για την ε, γνωμοδότηση όπως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονική. Για το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Keep voting. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε. 35 υπέρ, 2 κατά και μία αποχή συγχαρητήρια στον εισηγητή. So, thank you very much. I'm... Σας ευχαριστώ πολύ. Α, έχουμε κι άλλη. Έχουμε κι άλλη μη. Η προφορική. Μπλοκ στην ε, προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Φαίνεται ότι έχει εγκριθεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ. Κανένας κατά και καμία αποχή. Θα αναθέσω την Προεδρία τώρα στην Αρλίν, γιατί πρέπει να φύγω. Να μιλήσω με τον Πρόεδρο Μπούζεκ για την οικονομική διακυβέρνηση. Και γνωρίζω ότι ορισμένοι συγητές θέλουν να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Κάτι το οποίο και θα εκτελέσω. Όσοι είναι να φύγουν, να φύγουν ησύχως. Για να συνεχίσουμε με το, τις υποθέσεις του πρωινού. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση υποδήματα για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε 194 τροπολογίες. Νομίζω ότι η συγγήτρια ασχολήθηκε με μερικές από αυτές. Εν πάση περιπτώσει θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Ε, μπορείτε να συζητήσετε εκτός ε, αίθουσας, σας παρακαλώ. Γιατί θορυβείτε και επειδή έτσι και αλλιώς μας ακούνε μέσω διαδικτύου δεν είναι σκόπιμο να ακούγεται αυτός ο θόρυβος. Η κυρία Ποδηματά. Θα μιλήσω στα ελληνικά για να εξοικονομήσουμε χρόνο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους για τις 194 τροπολογίες ε, που λάβαμε ε, και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές και για τη συμβολή τους και για την ε, επικοδομητική συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Στη βάση των ε, τροπολογιών που λάβαμε έχουμε ήδη επεξεργαστεί μια σειρά από συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες στείλαμε σήμερα το πρωί στους σκιώδεις εισηγητές πριν μιλήσω για τις σημαντικότερες από αυτές τις συμβιβαστικές τροπολογίες, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις δύο βασικές παραμέτρους μέσω από τις οποίες, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσεγγίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα μέσα χρηματοδότησης. Η πρώτη παράμετρος είναι η συγκυρία την οποία διανύουμε. Μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, δύσκολη περίοδος για την Ευρώπη και ειδικά για την Ευρωζώνη, ίσως η πιο δύσκολη περίοδος από συστάσεως του ενιαίου νομίσματος, του ευρώ. Γνωρίζουμε όλοι ότι ανεξαρτήτως της ανάλυσής μας για το πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι δημοσιονομικές δυσκολίες και οι περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς θα έλεγα ακόμη και η πολύ σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την έγκριση του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού, όλα αυτά υποσκάπτουν σοβαρά, υπονομεύουν τις φιλόδοξες στρατηγικές και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα σε ορίζοντα δεκαετίας μέχρι το 2020 που γνωρίζουμε όλοι ότι αυτή θα είναι μια δεκαετία λιτότητας για τις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν σήμερα περισσότερο παραποτέ η αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, νέων πόρων, αποτελεί κατά τη γνώμη μου μονόδρομο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μέσα από τα προγράμματα λιτότητας, μέσα από τα προγράμματα αυστηρής δημοσιονομικής προσαρμογής είναι αυτοί που καλούνται να επομιστούν το κύριο βάρος του κόστους της κρίσης και γνωρίζουμε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι ότι υπάρχουν μαζικές διαδηλώσεις οι οποίες εξαπλώνονται απάκρου άκρου στην Ευρώπη και ότι επίσης το Ευρωβαρόμετρο δείχνει μια σημαντική αύξηση του ευρωσκεπτικισμού ακόμα και στους περισσότερο φιλοευρωπαϊκούς λαούς κατά παράδοση. Άρα λοιπόν η επιλογή που θα κάνουμε, το πόσο τολμηροί και φιλόδοξοι θα είμαστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στα μηνύματα που θα στείλουμε στους Ευρωπαίους πολίτες και στον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθεί η σχέση τους, η εμπιστοσύνη τους προς την Ευρώπη. Δηλαδή ότι πέρα από τα μέτρα λιτότητας, πέρα από τις περικοπές μισθών και συντάξεων, πέρα από τις αυξήσεις φόρων που έχουν κατά κύριο λόγο επίπτωση στους εργαζόμενους και στους καταναλωτές, η Ευρώπη μπορεί και θέλει να προτείνει, να δουλέψει πάνω σε εναλλακτικέ λύσεις που επιτρέπουν ένα δικαιότερο καταμερισμό. Έρχομαι τώρα στις ε, συμβιβαστικές τροπολογίες. Στο πρώτο κεφάλαιο, όπως ε, γνωρίζετε, μιλάμε για τη φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Εκεί ε, το κυρίαρχο ζήτημα είναι το θέμα της προώθησης ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε παγκόσμιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ήθελα σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι ε, πριν από δύο μήνες, στο πλαίσιο της υιοθέτησης της έκθεσης για την χρηματοπιστωτική, οικονομική ε, και κοινωνική κρίση, με μεγάλη πλειοψηφία και με στήριξη όλων σχεδόν των πολιτικών ε, ομάδων, υποστηρίξαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσεται υπέρ της επιβολής φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, τα έσοδα του οποίου θα βελτίωναν τη λειτουργία της αγοράς, μειώνοντας την κερδοσκοπία και θα συνέβαλαν στην χρηματοδότηση των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών και στη μείωση των δημόσιων ελλημάτων. Ε, το Κοινοβούλιο, σημειώνει η ίδια παράγραφος που υιοθετήσαμε πριν από δύο μήνες, θεωρεί ότι ο φόρος αυτός θα, έπρεπε, θα πρέπει να έχει την ευρύτερη δυνατή βάση, να υιοθετηθεί δηλαδή σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά ότι αν αυτό δεν συμβεί, ο φόρος θα πρέπει ε, να υιοθετηθεί καταρχάς στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασκήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα πίεση στο επίπεδο του G20. Και τέλος βεβαίως καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει γρήγορα μια μελέτη σκοπιμότητας ε, για να, ε, για να, μια μελέτη σκοπιμότητας λαμβάνοντας υπόψη ε, την διασφάλιση του δίκαιου επίπεδου ανταγωνισμού ανάμεσα στην ευρωπαϊκή αγορά και στις, και στις παγκόσμιες αγορές ε, να προχωρήσει λοιπόν τάχιστα στη μελέτη ε, μια τέτοια ε, μελέτη επιπτώσεων και στη συνέχεια να υποβάλει συγκεκριμένε νομοθετικέ προτάσει. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν έλλειψη συνέπεια απέναντι στην πλειοψηφία του Κοινοβουλίου που υπερψήφισε αυτή την παράγραφο, αλλά και η απουσία φιλόδοξων στόχων από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπό το φως των παρατηρήσεων που έκανα πριν, ε, εάν ε, ε, δύο μήνες μετά υποχωρήσουμε από αυτήν την διατύπωση που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης Μπέρευ. Στη βάση λοιπόν αυτών ακριβώς και αυτής ακριβώς της πρότασης στηρίζεται η συμβιβαστική τροπολογία της παραγράφου 7 που σας έχω στείλει σήμερα το πρωί. Ε, Περιτώ να επισημάνω ότι ασφαλώς και τασόμαστε υπέρ μιας παγκόσμιας συμφωνίας σε επίπεδο G20 δηλαδή καταρχήν. Αυτό καθίσταται σαφές στην στην έκθεση, αλλά ταυτοχρόνως πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ε, εθελοτυφλούμε, ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το, το momentum κινδυνεύει ε, να χαθεί και οι πιθανότητες για μια παγκόσμια συμφωνία στο ορατό μέλλον περιορίζονται. Άρα λοιπόν αν η Ευρώπη θέλει να αναλάβει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, ένα πρωταγωνιστικό ρόλο που της αντιστοιχεί ως της μεγαλύτερης χρηματοπιστωτικής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, θα πρέπει πιστεύω να πιέσει αποτελεσματικά ε, προχωρώντας την ενδελεχή μελέτη επιπτώσεων γύρω από αυτό το θέμα. Πέρα από το φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ε, οι συμβιβαστικές τροπολογίες που ε, έχουμε επεξεργαστεί και που σας μοίρασα σήμερα το πρωί, περιλαμβάνουν ασφαλώς και τις δύο κυριότερες επιπρόσθετες προτάσεις, δηλαδή την συνεισφορά των τραπεζών και τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, Ασφαλώς τα δύο αυτά εργαλεία πιστεύουμε ότι έχουν τη δική τους προστιθέμενη αξία. Ε, δεν πρέπει όμως να παραβλέψουμε ότι οι βάσεις φορολόγησης, τα έσοδα δηλαδή που μπορούν να προκύψουν και κυρίως ο ρόλος τον οποίο καλούνται να παίξουν τα δύο αυτά ε, χρηματοδοτικά εργαλεία είναι διαφορετικός από εκείνο που μπορεί να παίξει ο φόρος ε, επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και αυτή είναι μια παρατήρηση που αναγνωρίζεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από την τελευταία της ανακοίνωση για την φορολόγηση του χρηματοπιστωτικού τομέα όπου αναφέρει ε, ρητά ότι ο φόρος επί των ε, χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων δεν στοχεύει στην ίδια την συναλλαγή, ούτε στον τρόπο παραγωγής του κέρδους. Ε, ο φόρος επί των συναλλαγών στοχεύει, όπως είναι γνωστό, στην αντιμετώπιση των έντονα κερδοσκοπικών και μικρής διάρκειας συναλλαγών, και συνεπώς έχει μια επιπλέον προστιθέμενη αξία που αφορά στην διαφάνεια, στη σταθερότητα και στην αποτελεσματικότητα της χρηματοπιστωτικής ε, αγοράς. Ε, έρχομαι στο δεύτερο μεγάλο ζήτημα που, που περιλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση και που ε, αφορά στην παράγραφο που μιλάει για τα ευρωομόλογα και σε ό,τι αφορά την κοινή διαχείριση χρέους, τα Eurobonds και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση σημαντικών ευρωπαϊκών ε, υποδομών και σχεδίων, τα European Bond Projects. Στο δεύτερο αυτό σημείο διαπιστώνω ότι υπάρχει σημαντική σύγκληση από τις τροπολογίες ε, που έχουν υποβληθεί και ως εκ τούτου θα πω δύο λόγια κυρίως για το πρώτο θέμα, για τα ευρωομόλογα σε ό,τι αφορά ε, την κοινή διαχείριση μέρους του χρέους των κρατών μελών. Ε, η συμβιβαστική που προτείνεται σε αυτό το θέμα ζητά επί της ουσίας μια ε, ουσιαστική μελέτη επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, η οποία εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης και εν μέσω αναζήτησης τρόπων χρηματοδότησης μόνιμων μηχανισμών διαχείρισης κρίσης πιστεύω ότι δεν μπορεί να συνεχίσει ε, να αρνείται να εξετάσει τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου εργαλείου. Υπάρχουν διαφορετικές νόμες, υπάρχουν υποστηρικτές, υπάρχουν ε, αρκετοί που έχουν επιφυλάξεις. Ωστόσο θεωρώ ότι ε, σήμερα, και ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι να σας θυμίσω μάλλον ότι παρά τις αποφάσεις του ΕΚΟΦΗΝ και του Eurogroup την περασμένη Κυριακή το κόστος δανεισμού όχι πλέον μόνο των γνωστών αμαρτωλών ε, χωρών του Νότου, αλλά και άλλων χωρών όπως το Βέλγιο, όπως η Ιταλία. Το κόστος δανεισμού λοιπόν στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, τις μέρες που μιλάμε, ανεβαίνει σε ιστορικά ε, υψηλά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είχαμε χθε τον κύριο Τρισέ, δέχεται ε, κριτική από διάφορες πλευρές για την παράταση των προσωρινών μέτρων διασφάλισης της ρευστότητας. Λέω λοιπόν απλώς ότι είναι η κατάλληλη στιγμή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητήσει ε, μια ενδελεχή μελέτη επιπτώσεων ότι αξίζει τον κόπο ε, να μελετήσουμε σοβαρά ε, αυτή τη δυνατότητα ως ένα εργαλείο αναζήτησης μιας μόνιμης λύσης υπό αυστηρές προϋποθέσεις και στο πλαίσιο της συζήτησης και της διαπραγμάτευσης που διεξάγεται για τη νέα οικονομική αρχιτεκτονική στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο επίπεδο της Ευρωζώνης για την έκδοση ε, ευρωομολόγων. Τέλος, το τρίτο από τα μεγάλα ζητήματα, αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά στην αναθεώρηση που έχει ήδη ε, εξαγγελθεί από την πλευρά του Αρμόδιου Επιτρόπου, του κ. Σέμετα της, ε, της, της σημερινής ενεργειακής κοινοτικής νομοθεσίας. Πιστεύουμε ότι αυτή η αναθεώρηση πρέπει να γίνει με τρόπο που να περιλαμβάνει και τις εκπομπές άνθρακα, τις εκπομπές άνθρακα και το περιεχόμενο της ενέργειας, το ενεργειακό περιεχόμενο, ως βασικά κριτήρια της φορολογικής βάσης, καθώς με τον τρόπο αυτό θα ε, μια ε, ανισομερής αντιμετώπιση δραστηριοτήτων ε, ε, πολλών ετών που επιβαρύνουν τον περιβάλλον σε σχέση με εκείνες που δεν έχουν τέτοια συμπεριφορά και θα μπορέσουμε να μεταφέρουμε ένα τμήμα του φορολογικού άχθους από την εργασία όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα σε άλλες δράσεις. Η τροπολογία 167 ε, που ε, έχουν καταθέσει οι σκιώδεις, η συγκήτρια κυρία Χούπνερ και άλλοι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, νομίζω ότι αποτελεί μια ε, καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση και διαπραγμάτευση στο θέμα αυτό. Αυτά είχα να πω εισαγωγικά, κυρία Πρόεδρε, και για άλλη μια φορά ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για την συμβολή τους και για τις τροπολογίες τους. Uh, thank Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Πόδηματά. Θα συνεχίσουμε με, τον, με τους σκιώδεις και μετά τους ομιλητές. Η κυρία Χούμπνερ, ο σκιώδης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πόδηματά για το πολύ επικοδομητικό πλαίσιο συζήτησης όταν συζητήσαμε για πρώτη φορά ως σκιώδης. Ελπίζω να φτάσουμε σε συμβιβασμό στα περισσότερα ζητήματα τα οποία εντάσσονται στην έκθεση. Νομίζω ότι το καταφέραμε για τα περισσότερα ζητήματα, ίσως σε άλλα όχι. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της φορολόγησης του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια σε σχέση με τους όρους που διέπουν αυτό το φόρο. Για να ληφθεί δηλαδή μια τέτοια απόφαση και στο ε, Κοινοβούλιο, είμαστε διαχωρισμένοι. Υπάρχει μια μεγάλη διχογνωμία. Δεν είμαστε σίγουροι για την εισαγωγή αυτού του φόρου επί των ε, χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων ως βασικό όρο που να διέπει τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι εργάζεται σε μια μελέτη αντικτύπου, για μια μελέτη αντικτύπου, εάν εισαχθεί αυτός ο φόρος και θα περιμένουμε να δούμε την έκβαση αυτής της μελέτης αντικτύπου για να αποφασίσουμε για την εισαγωγή αυτού του φόρου, διότι μπαίνουμε σε εδάφη που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Υπάρχει και η εναλλακτική, αυτό το εναλλακτικό μέσο που αφορά τον φόρο δραστηριοτήτων. Δεν γνωρίζουμε και πολλά για αυτό το φόρο δραστηριοτήτων και όχι συναλλαγών και ευτυχώς αυτό είναι ένα ζήτημα που θα ενταχθεί στη μελέτη αντικτύπου της Κομισιόν. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα και από αυτά που μας είπε ο Επίτροπος σε ΜΕΤΑ ίσως ένα FAT, δηλαδή ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, ε, θα αποτιμηθεί από την ε, Κομισιόν το ταχύτερο δυνατόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να διαθέτουμε επαρκή χρόνο πριν λάβουμε τελική απόφαση, δηλαδή να δούμε τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου, πρωτίστως. Επίσης, επειδή, κυρία Πρόεδρε, μιλήσατε για τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Σάσεξ, θα ήθελα να πω ότι διάβασα αυτή τη μελέτη του Πανεπιστημίου του Σάσεξ και δεν είναι απόλυτα σίγουρη για το FTT, για τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Υπάρχουν ε, πολλές ε, αποκλίσεις απόψεων. Ε, υπάρχουν ε, χαμηλές δυνατότητες εσόδων πολλές φορές. Δηλαδή, ορισμένες μελέτες είναι πολύ, πολύ σαφείς ως προς αυτό. Δεν υπάρχουν δραστικές επιπτώσεις πάντα. Αυτή λοιπόν η αβεβαιότητα σε σχέση με τους όρους και τις επιπτώσεις του FTT υφίσταται μεταξύ εμπειρογνωμόνων. Και γι' αυτό και εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να το σκεφτούμε ως προς την τελική μας διατύπωση. Δηλαδή να καλύψουμε αυτή την αβεβαιότητα που υφίσταται. Ως προς τα ευρωμόλογα, υπήρξε μία γενική συνεννόηση σε σχέση με την ανάληψη υποχρεώσεων από την ΕΤΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με την ΕΤΕ για να δούμε κατά πόσο θα εισαχθεί αυτή το χρηματοπιστωτικό μέσο, πολιετές χρηματοπιστωτικό μέσο, μέσα στα πλαίσια των διαρθρωτικών μέτρων. Ως προς το δεύτερο κεφάλαιο, τμήμα του κεφαλαίου δηλαδή που αφορά τα ευρωομόλογα, νομίζω ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ρεαλιστές. Να δούμε δηλαδή τι μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια των διακλαδώσεων της παρούσας συνθήκης, ιδιαίτερα εάν επέλθουν μεγάλες αλλαγές επί της συνθήκης, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τα ευρωομόλογα. Η Επιτροπή όμως θα πρέπει να διερευνήσει ενδελεχώς τις δυνατότητες που διαγράφονται για να δούμε τι μπορεί να γίνει επί του θέματος και επίσης να δούμε τι μπορεί να γίνει μέσα στα πλαίσια της συνθήκης ή ε, αν αλλάξει κάπως η συνθήκη για να χρησιμοποιήσουμε ένα μέσο που χρησιμοποίησε και η Κομισιόν δυνάμει του άρθρου 143 της συνθήκης όταν είχε βοηθήσει με τα αυρομόλογα την Λετονία, την Ουγγαρία και την Ουγγαρία, καθώς και την, ε, την Λετωνία, την Ουγγαρία και την Πολωνία μέσα στα πλαίσια των χωρών που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά είχαν γίνει δυνάμει του άρθρου 143. Σε σχέση με την φορολόγηση του άνθρακα, δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτή την έκθεση. Εάν η Επιτροπή μας ταχθεί υπέρ αυτού, Ελπίζω να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στην ε, διαφορετική επίπτωση στα κράτη-μέλη, διότι ξέρουμε ότι υπάρχουν ομάδες κρατών μελών για τα οποία αυτός ο φόρος θα ήταν μεγάλη πρόκληση, ενώ για άλλες χώρες δεν θα σήμαινε τίποτα, δεν θα είχε σοβαρές επιπτώσεις. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά μετά την τελευταία μας συνάντηση με την κυρία Ποδήματα, είδαμε ότι φτάνουμε σε ένα συμβασμό ως προς αυτές τις παραγράφους, άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Γνωρίζω ότι δεν υπάρχει επαρκής χρόνος, αλλά προσβλέπω στις προτάσεις και τροπολογίες συμβιβασμού. Ελπίζω η συζήτηση να είναι επικοδομητική όπως ήταν μέχρι τούδε για τα περισσότερα ε, ζητήματα τα οποία παραμένουν επιτάπητος και δεν έχουν ε, διασαφινιστεί επαρκώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Εγώ δεν ζήτησα το να μιλήσω στη συζήτηση αυτή αλλά και δεν θέλω να κάνω μια διμερή συζήτηση μαζί σας κυρία Χιούμπνερ αλλά οφείλω να πω ότι δεν μπορείτε να παρουσιάσετε την έκθεση με τέτοιο τόσο αρνητικά Λέγεται ε, στην έκθεση, η οποία είναι πολύ ε, καλή κατά την άποψή μου και λέγεται ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε ορισμένα πράγματα και στο εξωτερικό εμπόριο. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι το θέμα βέβαια επιτρέπεται δηλαδή μπορεί να γίνει και λέγεται και αυτό εδώ το θέμα βέβαια είναι αν μας αρέσει, αν θέλουμε να το κάνουμε ή όχι. Λάμπερτ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαρι... και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι Ντανούτα Βιμπνελ. Θα ήθελα να απαντήσω. Δεν θα μιλήσω υπέρ κατά του τη... Έχει γίνει αρκετή κουβέντα γι' αυτό. Για το φόρο. Αλλά όπως είπες Ντανούτα, υπάρχει αβεβαιότητα ε, δεν έχουμε όλες τις, ε, όλα τα στοιχεία. Εγώ προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα και το management στον ιδιωτικό τομέα παίρνει αποφάσεις ακόμη και υπό αβέβαιες συνθήκες. Ε, με συνέστηση ότι τα πράγματα είναι ρευστά, το management παίρνει αποφάσεις. Αυτό καλείται να κάνει. Οι αποφάσεις που παίρνονται τώρα παίρνονται χωρίς να έχει γίνει πλήρης ανάλυση του αντικτύπου, χωρίς να έχουν γίνει πλήρης ανάλυση. Όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση ή άλλες κυβερνήσεις έδωσε απεριόριστες εγγυήσεις στις τράπεζες, δεν ήξερε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος αυτής της κίνησης. Και τώρα βεβαίως Λυπούμεθα γι' αυτό. Πολλά κράτη-μέλη αποφάσισαν να, ε, να μειώσουν τα ελλείμματά τους ε, επεμβαίνοντας στην πλευρά των δαπανών. αλλά χωρίς να κάνει προηγούμενα μελέτη. Ε, εγώ αν ήμουν σοσιαλιστής, γιατί οι περισσότεροι σοσιαλιστές χώρες κάνουν αυτό. Ε, θα το πρόσεχα ιδιαίτερα, διότι ε, μεγαλώνουμε το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών με αυτόν τον τρόπο. Διότι δεν, δεν έχει γίνει οικονομική ανάλυση. only place. But so if you believe that αν πιστεύετε όμως ότι οι κυβερνήσεις έχουν κάποια πράγματα να κάνουν, θα πρέπει να κάνουν ορισμένα πράγματα, να αναζητήσουν, να κοιτάξουν την πλευρά των εσόδων, να αναζητήσουν καινούριε πηγές. Αλλά αυτό να το κάνουν μετά από πλήρη ανάλυση. Μια πηγή θα ήταν ο τόξος αυτό, ο τόκος, ο φόρος αυτός. Αυτή τη στιγμή η κύρια πηγή είναι η εργαζόμενη. Και πραγματικά δεν έχει γίνει ανάλυση για όλες τις δυνατές πηγές αλλά κάποια απόφαση πρέπει να πάρθει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ονείως για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Ε? Θα πρέπει να πάρετε μια απόφαση παρόλο που δεν έχουμε την πλήρη εικόνα ή την πλήρη, την πλήρη ανάλυση. Να ενσωματώσουμε στην απόφαση που θα πάρουμε το ρίσκο που παίρνουμε χωρίς να έχουμε όλα τα στοιχεία. Γιατί ο χρόνος περνάει και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να κοιτάξουμε τις δαπάνε καθόλου, αλλά για την πλευρά των εσόδων πρέπει να προχωρήσουμε έτσι όπως είπα. Τώρα για το ευρωμόλογα πάλι τα πράγματα είναι ρευστά. Ορισμένοι λένε ότι μπορούμε να κάνουμε μεγάλα κέρδη με τα ευρωομόλογα. Μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά και πάλι δεν έχουν μελετηθεί τα πράγματα. Όταν αρχίσαμε να επιτρέπουμε τις συναλλαγές με, παράλογο, με παράγωγα, <laughs> συγγνώμη, ε, δεν ξέραμε τι θα γινόταν. Για πολύ σοβαρούς οικονομικούς λόγους χρησιμοποιούν τα παράγωγα κάποιοι τα χρησιμοποιούν σαν εργαλείο για να προστατευτούν, αλλά υπάρχουν και οι άλλοι που τα χρησιμοποιούν για κερδοσκοπικό σκοπό. Λοιπόν, για αυτούς που τα χρησιμοποιούν σωστά, για προστασία, να προστατεύσουν ορισμένα πράγματα, ε, δεν θα πρέπει να τους βοηθήσουμε. Επειδή υπάρχουν και άλλοι κερδοσκόποι, θα πρέπει να σταματήσουμε τα πράγματα. Ξέρουμε ότι έχουμε ένα εργαλείο, το οποίο ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει κατάχρησή του, αλλά το διατηρούμε. Το ίδιο θα γίνει και με τα ευρωομόλογα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να τους μηδενίσουμε. Αν πούμε θέλουμε μηδέν ρίσκο, αυτό σημαίνει μηδέν ομόλογα, ευρωομόλογα. Δεν μπορεί να πάρθει απόφαση για τα ευρωομόλογα. Αν πούμε ότι ή τα πλεονεκτήματα του F, του, του, υπάρχουν πλέον εκτίματα στα ευρωομόλογα, ε, τότε πρέπει να αναλάβεις και το ρίσκο. Okay, Mr. Ο κύριος Χάγκλαντ, εκ μέρους της ομάδας σας παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριος Σμιθ ε, σήμερα είναι στο Κονγκό, είναι σκιώδης και έτσι έχω την ε, ευκαιρία και την τιμή θα πάρω το λόγο εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω για την έκθεση και για τις συμβαστικές προτάσεις που γίναν. Θα ήθελα να πω ότι από πολιτικής απόψεως η κατάσταση είναι τουλάχιστον προκλητική. Βεβαίω υπάρχει η συζήτηση των ιδίων πόρων, ε, η οποία είναι σημαντική αν θέλουμε ιδίους πόρους ή όχι. Όμως συγχρόνως την ομάδα μας είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε πλήρεις αναλύσεις ούτως ώστε όταν προτείνουμε κάτι να είναι εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό. Για την πρόταση τώρα κάποιων φόρων Ίσως είναι δύσκολο να κάνει κανείς προτάσεις αυτές αν δεν έχει γίνει πλήρης η ανάλυση. Αλλά επειδή είπαμε ότι πρέπει να γίνουν και φιλόδοξες προτάξεις για τους ίδιους πόρους αλλά και για το, το φόρο αυτό των συναλλαγών, ε, καλώς ας... Ε, γίνει και η πρόταση για τον ευθύτη. Από την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να έχουμε και κάποια υπομονή, να περιμένουμε λιγάκι, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μπορεί να τρομάξουμε και ορισμένους ανθρώπους. Αν πιώσουμε, για αν προωθήσουμε και για ιδεολογικούς λόγους υπερβολικά τον φόρο αυτό, μπορεί να κάνουμε λάθη. Υπάρχουν επιχειρήματα και υπέρ και κατά του φόρου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το καλοκαίρι ήταν τελείως επικριτικό για το φόρο αυτό. έχουμε έναν εταίρο, κύριο και μεγάλο εταίρο που μιλάει υπέρ της διάσωσης των χωρών από τη μια, αλλά και είναι και κατά του φόρου αυτού από την άλλη. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάρουμε, μπορέσουμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και να μην προτρέχουμε να μην προσπαθούμε να προωθήσουμε πράγματα για ιδεολογικούς λόγους αν δεν έχει γίνει πλήρης οικονομική ανάλυση τους και ανάλυση αντικτύπου. Ξέρουμε ότι πολλές από τις οικονομικές δραστηριότητες του Λονδίνου μετακομίζουν στην Ελβετία ε, φοβόμαστε ότι κάποια πράγματα που ε, προτείνονται στην έκθεση μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και άρα να πληγώσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέω ότι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο και να υπάρχουν και επιτυχίες. Αλλά ε, Θέλω να πω ότι όλα αυτά έχουν αντικτύπους, επηρεάζουν τα πάντα τα πάντα, ε, πειράζουν τους ίδιους πόρους, οπότε δεν θα πρέπει να βιαστούμε διότι τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν για όλους τελικά. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ludwigson. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτή την έκθεση θα πρέπει να έχουμε τις λεπτές χρειές και τη σωστή ισορροπία. Υπάρχουν λυπείς γνώσεις στον τομέα τον οποίο πραγματευόμαστε. Υπάρχουν ε, υποσχέσεις σε σχέση με τις νέες μεθόδους χρηματοδότησης, πλην όμως δεν έχουμε σαφή εικόνα ε, σχετικά με την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα περνάμε ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και θα έπρεπε να τους πούμε ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό έρισμα γνώσεων, το ταχύτερο δυνατόν για να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να εντατικοποιήσει τι εργασίε για να ε, εκπληρωθούν οι υποσχέσει σχετικά με το φόρο των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Για αυτό το φόρο, όταν κάνουμε την ανάλυση των συνεπειών, ε, θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε τον διάλογο, αλλά να γίνει πιο συγκεκριμένο ο διάλογος, να γίνει ευρεία διαβούλευση με τι εταιρείε, του πολίτες, να ξέρουμε για ποιο ακριβώς στόχο θα χρησιμοποιηθεί αυτός ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ε, και θεωρώ ότι δεν είναι ακόμη αρκετά διαρθρωμένη η πρόταση περί φόρου. Θα έπρεπε επίσης ε, να κάνουμε μια ευρύτατη ανάλυση για το νέο φόρο σχετικά με την ε, δομή των ίδιων των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε στα γενικότερα συμφραζόμενα αυτόν τον φόρο πώς θα λειτουργήσει επίσης. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι το σουηδικό παράδειγμα προβάλλεται μέσα στις τροπολογίες που υποβάλαμε και εφαρμόζεται και τη δεκαετία του 80 αυτός ο Σουηδικός φόρος ε, και δεν ευωδόθηκε. Οπότε θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Τώρα βέβαια αυτός ο φόρος, ο σημερινός που συζητάμε τώρα, διαφέρει από τον σουηδικό φόρο. Ε, ε, και ποια είναι η διαφορά, ότι ήταν 20 έως 100 φορές υψηλότερος αυτός ο φόρος. Άλλη διαφορά, ε, ε, κάλυπτε μόνο ένα κομμάτι της αγοράς αυτός ο σουηδικός φόρος, ενώ τώρα θα θεωρείται ως γενικευμένος κανόνας. Ε, θα πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε τα συμπεράσματα, αλλά να μην απλοποιούμε την κατάσταση. Το σουηδικό παράδειγμα Πάντω ε, μας δείχνει ότι πρέπει να έχουμε κάποιους ενδιασμού σε σχέση με το, τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει ένας τέτοιος φόρος. Ε, μην ξεχνάτε επίσης πώς λειτουργούσαν τα κινητά τηλέφωνα το, τη δεκαετία του 80. Υπήρχαν περιορισμοί τότε. Όμω τώρα με τις τεχνολογικέ εξελίξεις υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες στον τομέα τη κινητής τηλεφωνίας. Ελπίζω το ίδιο θα συμβεί και με του φόρου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Χεκμάρκ ε, και να σας πω ποιοι άλλοι είναι στον κατάλογο. Κύριε Λάμπερ, συντομία και μετά θα δώσουμε το λόγο στην ε, κυρία Ποδηματά. Α, δεν είχατε ξαναζητήσει το λόγο. Δεν πειράζει. Ο κύριος Χέκμαρκ, σας ευχαριστώ. Ε, πρώτα απ' όλα σε σχέση με τις ε, συζητήσεις που έγιναν για τα ευρωομόλογα. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε την κατάσταση, διότι... Ε, θα πρέπει να συνδέσουμε αυτή τη συζήτηση με τη συζήτηση για την διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ. Ε, δηλαδή συζητάμε για την, ε, το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων. Ε, συζητούμε για τα υπερβολικά ελλείμματα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταργήσουμε την ε, de facto ύπαρξη των στοιχείων που γνωρίζουμε ήδη στο τωρινό οικονομικό περιβάλλον, να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και διαπιστώνω διάφορα προβλήματα με το ενδεχόμενο ε, εφαρμογή των ευρωομολόγων. Τα τα ίδια τα ευρωομόλογα, όχι γενικότερα τα προγράμματα που καλύπτουν τα ευρωομόλογα, δεν νομίζω ότι θα μας οδηγήσουν σε επιτυχία αν θέλουμε να ε, προοδεύσουν τα ευρωπαϊκά το, να, συγγνώμη, να προοδεύσει το ευρωπαϊκό νόμισμα γενικότερα. Τώρα για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έχω ξαναπεί αυτά σε προηγούμενες συζητήσεις, είχα τονίσει κάτι που κατεμένει πάρα πολύ σημαντικό τι θα συμβεί αν έχετε έναν ειδικό φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όπως είπε και ο κύριος λάμπες χρειαζόμαστε ε, κάποιο φόρο και μπορεί μάλιστα να είναι και αρκετά καλή αυτή η φόρη. Βεβαίως, αλλά αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να αντικατευθύνουμε κατευθύνουμε προς την εξέταση των στόχων που επιδιώκουμε για να μειώσουμε την κερδοσκοπία παραδείγματο χάρη μάλιστα αλλά είναι δύσκολο να ορίσουμε την ε, κερδοσκοπία γιατί δείτε πόσοι αντιμετωπίζουν δημοσιονομική κρίση ε, Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία ε, βέβαια όταν δανείζονται κάποιοι ούτως ή άλλως διατρέχουν κάποιο κίνδυνο και νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι περί του ότι ε, θέλουμε να μπορούν να δανειστούν αυτές οι χώρες. Θέλουμε να διατρέξουν αυτό το κίνδυνο εφόσον χρειάζονται δάνειο. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση αν επιβάλλουμε επιπλέον ένα φόρο πέρα δηλαδή από το κίνδυνο που θα διατρέχουν οι χώρες. Διότι πρέπει να έχουμε επίγνωση του ότι αυτοί που θα καταβάλουν αυτό το φόρο είναι οι ίδιοι που δανείζονται χρήματα δεν υπάρχουν δωρεάν χρήματα κρυμμένα μέσα σε κάποιο υπόγειο στην Ευρώπη που ε, θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στα Σουηδικά ε, ε, θα προσπαθήσω, έχουμε μία παροιμία και θα προσπαθήσω να τη μεταφράσω ή μάλλον. Τέλο πάντων, το νόημα είναι ότι άμα συνδυάσετε όλα τα υφιστάμενα στοιχεία μπορείτε να εκπληρώσετε το όνειρό σας για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών εννοώ ότι πρέπει να διευκρινίσουμε κατά ποιο τρόπο ακριβώς επικουρούμε τις χώρες και τις περιοχές του κόσμου που χρειάζονται κεφάλαια ε, επιβάλλοντας φόρο επί των κεφαλαίων που αναμένεται ε, αυτές οι χώρες να δανειστούν. Ο στόχος είναι να μειώσουμε τις βραχυπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Μάλιστα. Πρέπει να συμφωνήσουμε όμως ότι είναι κακέ εισαγωγικά αυτές οι βραχυπρόθεσμε συναλλαγέ. Αν δεν επιβάλλουμε φόρο σε αυτές τις ε, ε, συναλλαγές, όλες αυτές οι χώρες θα βυθιστούν ακόμη βαθύτερα στην κρίση, γιατί μόνο λίγες ε, θα χαρούν να δανειστούν μακροπρόθεσμα για να χρηματοδοτήσουν ολόκληρο το έλλειμμα τους, χωρίς όμως να τους δίνει τη δυνατότητα να προβούν σε βραχυπρόθεσμες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αν, ε, αν τώρα συζητάμε αν θα είναι αποτελεσματικός αυτός ο φόρος των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ποιο είναι ο στόχος να μειωθεί ο αριθμός των βραχυπρόθεσμων ε, ε, πράξεων και η διόγκωση των προβλημάτων σε όλες αυτές τις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, ο συνάδελφος μου, ο κύριος Λούντβικσον, ε, είπε ότι η πρώτη απόπειρα ήταν αποτυχία και τώρα θα πρέπει να το ξαναπροσπαθήσουμε. Θαραλέο τον βρίσκω. Δεν θέλει να σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ε, αλλά θα συνδυάσω την απάντησή μου με την επιχειρηματολογία του κύριου Λάμπερς. Είπατε ότι χρειαζόμαστε ε, τέτοιους φόρους. Ξέρετε τι έγινε. Η Σουηδία τότε, εκείνη την περίοδο, είχε τον υψηλότερο φόρο εισοδήματος ε, και εισαγάγαμε τον φόρο Τόμπιτ, έτσι λεγόταν τότε. Ήταν φόρος επιχρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών. Περί αυτού ε, είναι ο λόγος και τώρα. Αλλά τι έγινε, ε, το μεγαλύτερο μέρος ε, των εμπορικών συναλλαγών που πήγανε στο Λονδίνο. Ε, εκεί χάρηκαν βέβαια με αυτή την ιστορία, αλλά δυστυχώς ε, στη Σουηδία δεν είχαμε αυξημένα φορολογικά έσοδα. Ε, χάσαμε πολύ περισσότερα από τα έσοδα που λάβαμε. Πολλοί μετακο... δεν μετακόμισαν στην... στο Λονδίνο παρότι είχαμε τον υψηλότερο φόρο εισοδήματος. Οι συναλλαγές πήγαν στο Λονδίνο, όχι οι άνθρωποι, γιατί οι συναλλαγές είναι φορητές. Και αν θέλετε μάλλον δεν καταλαβαίνω γιατί θέλει το Δήμορο στη Σανγκάη να γίνει ο πιο ευτυχής άνθρωπος ε, του κόσμου. Δηλαδή, αυτό θα συμβεί αν επιβάλλουμε φόρο χρηματοπιστωτικά ε, συναλλαγών στην Ευρώπη. Θα πάνε συναλλαγέ αλλού στην Ευρώπη και κυρίως σε χώρε όπως η Κίνα. Ε, συγκεκριμένα στη Σανγκάη θα πάνε συναλλαγές. Όπως είπε και ο κύριος Λούτβικσον, ήταν αποτυχία αυτός ε, ο φόρος ε, τη δεκαετία του 80 όταν εφήβραμε το φόρο γιατί πήγαν οι συναλλαγές στο Λονδίνο. Μα κανείς δεν διαφωνεί για αυτά τα συμπεράσματα. Τώρα μας λέει ο κύριος Λούτβικσον ότι έχουμε μετεξελίξει το όπλο αυτό και είναι πιο εξελιγμένο και άρα πιο αποτελεσματικό. Μάλιστα. σίγουρα δεν θα πάνε οι, οι συναλλαγές στην Ευρώπη, θα πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου. Αυτή θα είναι η διαφορά. Ξέρω επίσης ότι συζητάμε για την ανάγκη ε, ε, διεξαγωγής ε, αξιολόγηση αντικτύπου. Ναι, αλλά πριν προτείνουμε το φόρο να κάνουμε την αξιολόγηση αντικτύπου, να ξέρουμε. ο η εισηγήτριά μας ε, που άρχισε αυτή τη συζήτηση δεν έδειξε και ούτε και ο κύριος Λάμπερ στην παρέμβασή του μας έδειξε για ποιο λόγο αυτές οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, ε, ο φόρος μάλλον επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών θα ε, μειώσει την κερδοσκοπία και δεν θα παρεμποδίσει, δεν θα παρακολουθήσει τις εμπορικές συναλλαγές. Ναι, το αντίστροφο ισχύει, κατά τη γνώμη μου. Οι χρηματοπιστωτικές ε, συναλλαγές. Ε, μάλλον αυτό που μα ενδιαφέρει είναι η μείωση της ε, κερδοσκοπίας. Αυτό ο κίνδυνο που ε, διατρέχουμε είναι να μειωθούν οι επενδύσει και οι πραγματικέ εμπορικέ συναλλαγέ και θα εμποδίσουμε την ανάπτυξη φτωχότερες περιοχές του κόσμου και θα διωγγώσουμε τα δημοσιονομικά έλλειμμα. Δεν καταλαβαίνω ε, με ποιο ακριβώ τρόπο θα αναβαθμιστεί η κατάσταση με αυτό το φόρο. Μάλιστα σα ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικέ οι παρατηρήσει και πολύ ενδιαφέρον ε, είναι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να γίνει αξιολόγηση αντικτύπου, οπότε συμφωνεί μαζί σα, κυρία Φόρτ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη ε, εξ ονόματος ε, της Κιόδους που δεν ε, μπόρεσε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Σε σχέση με ορισμένες τροπολογίες που πρότεινε ο συνάδελφος. Φαινόμαστε ασυνεπείς ως προς το μήνυμα που αποστέλουμε με αυτό το έγγραφο έναντι του μηνύματος που αποστέλουμε στα κράτη-μέλη ως προς το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης διανύουμε δύσκολους καιρούς με μία αγορά που κλειδονίζεται με spreads τα οποία γνωρίζουν πολύ μεγάλες αυξομοιώσεις και στο έγγραφο περί οικονομικής διακυβέρνησης αρχίζουμε λέγοντας ότι πρέπει να έχουμε προληπτική φορολογική πολιτική και η προληπτική φορολογική πολιτική βασίζεται σε μακροοικονομικούς συντελεστές και με, βασίζεται σε δοκιμές αντοχής. Τι θα κάνει αυτή η φορολόγηση στον επιχειρηματικό κόσμο. Πώς συσχετίζονται τα δύο είχαμε εμπειρογνώμονες που μας είπαν τη Δευτέρα τι έγινε στην Ιρλανδία. Δηλαδή βασιστήκαμε στη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας και όταν χάθηκε η αγορά ακινήτων χάθηκε και αυτή η πηγή εσόδων. Άρα δεν είναι συνετό να έχουμε φορολογικό προγραμματισμό χωρίς ε, να έχουμε μία μελέτη που κύριε Λάμπερτς. Βεβαίως δεν υπάρχει βεβαιότητα 100% κύριε Λάμπερτς, αλλά, αλλά μην ε, κάνουμε ένα άλμα μέσα σε μαύρες τρύπες χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνουν. Γιατί αυτό που λέμε ότι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη πρέπει να το κάνουμε και εμείς. Τα χρήματα, τα έσοδα από τη φορολογία δεν ε, είναι κάτι το αυτονόητο. Και δεν μεγαλώνουν στα δέντρα αυτά τα έσοδα. Δεν είναι μια ανεξάντλητη πηγή και από όσο γνωρίζουμε υπάρχει μεγάλος άλληλος συσχετισμός μεταξύ προϋπολογισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα έσοδα για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να έχει αυτό αντίκτυπο στα κράτη-μέλη. ως προς τον φόρο ε, χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, είναι πολύ δύσκολο για ορισμένα κράτη-μέλη να εισαγάγουν ε, έναν τραπεζικό φόρο. Εμείς στη χώρα μου το κάναμε, άλλοι όμως αποφάσισαν να μην το κάνουν, πέρα από το σχέδιο διάσωσης. Και μία από τις τροπολογίες που υποβάλαμε υπενθυμίζει ότι αυτός ο φόρος θα δοθεί στο κοινό για αυτό που έδωσαν για τη διάσωση των τραπεζών. Θα επιστραφεί δηλαδή στο κοινό. Ως προς τα ευρωομόλογα, στο πακέτο οικονομικής διαχείρισης, διακυβέρνησης, τονίζουμε ότι ε, οι φούσκες αυτές αφορούν μια γενικότερη διαδικασία ε, ζημίας και τα ευρωμόλογα, αν τα χρησιμοποιήσουμε ως μόχλευση δυνάμει της ΕΤΕ, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτή τη ζημιογόνο κατάσταση. Άρα θα θέλαμε να πούμε ότι υπάρχουν ε, καλή τρόπη μόχλευσης δημόσιου και ιδιωτικού χρήματος. Συμφωνούμε απόλυτα ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές δεν μπορούμε να έχουμε χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό θα βασιστούμε στο δημόσιο. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα όρια κινδύνου. Διαφορετικά προσκρούμε στα προβλήματα που είδαμε σε ορισμένα κράτη-μέλη. Εμείς λέμε ας δούμε αυτή την οριοθέτηση μέσα στα πλαίσια της δημόσιας λογοδοσίας. Ο κύριος Μπούλμαν. Ο συνάδελφος Χουκμακ είπε ότι είναι πιο λογικό οι μελέτες για τους η αξιολόγηση αντικτύπου να γίνεται πριν να πάρθει κάποια απόφαση. Γι' αυτό ζητήσαμε το Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια μελέτη. Ήσαμε τώρα όμως, Δεκέμβρη 2010, δεν έκανε τη μελέτη αυτή η Κομισιόν. Πέρασαν τρία τέταρτα της χρονιάς και δεν υπήρξε καμία κίνηση στο θέμα αυτό. Και γι' αυτό φταίει η Κομισιόν. Εδώ όμως σταματώ να συμφωνώ. Θα ήθελα να πω στον κύριο Χίμπνερ ε, και άλλους συναδέλφους το εξής. Με... Προσπαθώ να είμαι φιλικός και ευγενικός, αλλά είμαι υποχρεωμένος να πω ότι δεν πιστεύω πως έχετε σοβαρή συνέστηση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, η Ευρωζώνη. Δεν πήρατε σε σοβαρά το επιχείρημα που ανέφερε ο κύριος Λάμπερτ ότι η οποιαδήποτε απόφαση παρθεί τώρα στο, για το α θέμα επηρεάζει και άλλες αποφάσεις για χίλια δυο άλλα θέματα. Η κατάσταση στην οποία ζούμε είναι πολύ σοβαρή. Αν προσθεθεί και άλλο ένα μεγάλο κράτος μέλος στη, στις χώρες που χρειάζονται σωτηρία από την Ευρώπη, τότε τα 750 δις του μηχανισμού κλείνουν, τελειώνουν. Ξέρετε πολύ καλά λοιπόν πόσο ή μάλλον πρέπει να, να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και να συνειδητοποιήσετε ότι αν κάποια άλλη χώρα και μη μεγάλη χώρα βρεθεί στην ίδια κατάσταση με την Ελλάδα και την Ιρλανδία τα πράγματα είναι ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα τραγικά για την Ευρωζώνη. Ξέρετε τι γίνεται στις διάφορες χώρες. Ξέρετε τι έχει γίνει με τους προϋπολογισμούς των περισσότερων χωρών. Ξέρετε πώς θα επηρεάσει τις χώρες σαν την Ελλάδα και την Ιρλανδία, οποιαδήποτε κίνηση εδώ. Τι γίνεται με τις εξαγωγές, εισαγωγές. Υπάρχουν άλλες χώρες που δεν μπορούν να καλύψουν τη ζήτησή τους ή που δεν θα μπορούν να καλύψουν εσωτερική του ζήτηση ε, αν συμβούν ορισμένα πράγματα και πουθενά μα πουθενά δεν υπάρχει καμιά εγγύηση για το ότι η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να υφίσταται σε δέκα χρόνια θέλουμε η ενιαία εσωτερική αγορά και η Ευρωζώνη να επιβιώσει και να ε, ναι, δυναμώσει. Θέλουμε νέα, νέες χώρες στην Ευρωζώνη ε, στο μέλλον. Αλλά δεν υπάρχει καμιά εγγύηση, επαναλαμβάνω, καμία εγγύηση για το ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα πράγματα αυτά σε δέκα χρόνια. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Γι' αυτό πρέπει να καθίσουμε, να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά πού βρίσκονται οι πηγές από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μία ανάκαμψη. Και αυτό αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουμε. Πρέπει να την πάρετε. Η έκθεση της συναδέλφου Ποδηματά δεν θα είναι μια οποιαδήποτε έκθεση στην Ολομένια ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα είναι η έκθεση κατά τη συζήτηση της οποίας οι πολιτικές ομάδες θα πάρουν θέση γι' αυτό το θεμελιώδες δίλημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί ο καθένας μας θα ρωτηθεί, εσείς θα ρωτηθείτε από την ποια από ποια πλευρά στεκόσαστε για το θέμα αυτό αν μπλοκάρετε ή δεν μπλοκάρετε ξέρετε πολύ καλά ε, ότι οι φόροι ε, συλλέγονται από τα κράτη-μέλη. Εκείνο που γυρεύουμε αυτή τη στιγμή είναι από την Κομισιόν να κάνει μια πρόταση, έτσι, από την ψηφοφορία και την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέχρι όταν αρχίσουν να εφαρμόζονται πολύ συγκεκριμένα κάποια πράγματα θα περάσει πολύ καιρός θα κυλήσει πολύ νερό στα βλάκια αλλά αν δεν δώσουμε αυτό το ελάχιστο μικρό μήνυμα δεν έχουμε κάνει τίποτα αυτό τώρα ρώτησε ο συνάδελφος τι θα γίνει μέχρι του χρόνου του Γενάρη για το economic governance. Πάρα πολύ <coughs> σημαντικό είναι το ερώτημα αυτό. Είναι για τον επόμενο Ιούνιο, αλλά τώρα καλούμεθα να δώσουμε απάντηση και να στείλουμε ένα μήνυμα για τα ερωτήματα που υπάρχουν κύριοι. Συγγνώμη, αλλά δεν τελειώνει η συζήτηση για τα πολύ σοβαρά αυτά θέματα εδώ. Κύριος Γκοζές. Εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορεί κάποιο να είναι από τη δεξιά, από την κέντρο δεξιά, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε και τυφλοί ούτε μουγκοί. Αυτό που έγινε στην κρίση και δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε και να προσποιηθούμε ότι όλα είναι όπως πριν γιατί οι τράπεζες έχουν αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δανείων που ε, συνήθηκαν και μπορούν τώρα άνετα να προχωρήσουν. Δεν σύμφωνα με τον κύριο Πουλμαν όταν μας λέει ότι μέσα από αυτή την έκθεση ε, θα ε, ε, μετρήσουμε τις δυνάμεις των μεν και των δε. Όχι, το 2010 το είχαμε πει, κανείς δεν μας άκουσε όμως και και το 2015 πάλι δεν θα λαμβάνεται υπόψη η έκθεση. Θα μπει σε ένα σιρτάρι ε, και θα είναι σκονισμένη. Αυτό που είναι σημαντικό να γίνει σήμερα είναι με ρεαλιστικό τρόπο να εντοπίσουμε ποια στοιχεία μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε. Τι ε, να πρεσβεύουμε τέτοιε μεγάλε ιδέε δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν. Εδώ εκπροσωπούμε του πολίτε και όπω ε, και εσεί συζητώ με τους πολίτες, ξέρω για ποια πράγματα ανησυχούν και το πρόβλημα των πολιτών δεν είναι να μάθουν να πάνε καλά τα πράγματα στη City ε, του Λονδίνου. Το θέμα είναι να ε, τα χρηματοπιστωτικά ποια κατεύθυνση θα ε, ακολουθήσουν, θα εξυπηρετήσουν την πραγματική οικονομία ή όχι, θα είναι χρήσιμα για τα δημόσια οικονομικά ή όχι. Να οι πραγματικές ερωτήσεις, επ' αυτών πρέπει να προβληματιστούμε. δεν πρέπει να ε, ε, τοποθετούμαστε δογματικά για αυτά τα ζητήματα. Ωραία, σήμερα μας λένε να κάνουμε αξιολόγηση αντικτύπου. Πολύ ωραία, συμφωνώ. Όμως, έχω την εντύπωση σήμερα ότι συχνά η αξιολόγηση αντικτύπου, όπως είπε σωστά ο κύριος Λάμπερτς, ε, είναι ένας τρόπος για να συγχέονται όλα και να μπερδεύουμε τον κόσμο όταν σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία παραδείγματο χάρη, όταν καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία και ποτέ δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στοιχεία στη διάθεσή μα, γιατί υπάρχουν απρόβλεπτοι παράγοντε, υπάρχουν μη μετρήσιμα στοιχεία που έχουν ω αποτέλεσμα ε, μία απόφαση που λαμβάνεται σε ένα, μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι καλή ή κακή και σε κάποια άλλη χρονική στιγμή αλλάζουν τα δεδομένα. Ε, Ε, οφείλουμε να αναρωτηθούμε αν ε, χρειάζεται αυτός ο φόρος. Επί της αρχής να αναρωτηθούμε, όπως σας παραπέμπω και στην έκθεση της κυρίας Περβάνσε, ε, ε, ε νομίζω ότι στην πράξη πρέπει να αναρωτηθούμε και για τη φορολογική βάση αλλά κυρίως για τη χρησιμοποίηση, τη χρήση, τη μελλοντική χρήση αυτού του φόρου για τα ε, χρηματοπιστωτικά θα επαναλάβω κάτι που σας είπα ε, εσχάτως. Ε, σκανδαλίστηκα και τονίζω τον όρο που χρησιμοποιώ ε, όταν είδα τις αντιδράσεις κάποιων εναλλακτικών ε, επενδυτικών κεφαλαίων, κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδυνού, τα hedge funds, μόλις είδαν ότι εγκρίθηκε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου. Μας είπανε μάθα να τηνάξετε τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία, θα βυθίσετε ακόμη περισσότερο στην κρίση φτωχότερες χώρες. Θα σκοτώσετε την οικονομία αν ε, εφαρμοστεί το ψήφισμα. Και τελικά ε, με το ψήφισμά μας θεώρησαν ότι δεν ρυθμίσαμε τίποτα. Μα άδικο έχουν γιατί δεν έχουν την οδηγία και υπάρχει και η ρήτρα ενδιάμεσης αναθεώρηση σε τρία χρόνια. Οι περισσότεροι εδώ θα είμαστε και δεν θα ε, ξεχάσουμε με ποιο τρόπο προσπάθησαν να μας κοροϊδέψουν. Νομίζω ότι χρειάζεται συλλογικό προβληματισμό και όχι κομματικό. Όχι να λέμε εγώ θέλω αυτό, εκείνο, βάλε αυτό, βγάλε αυτό. Ε, νομίζω ε, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε εκτελεστικό όργανο. Εμείς πρέπει να κάνουμε εισηγήσεις, να ε, φέρουμε ναι, καινούργιες ιδέες για να σημειωθεί η πρόοδος ε, και να ρίξουμε την μπάλα πέρα από το σημείο που θέλουμε να προσγειωθεί. Ο κύριος Λάμπες ευχαριστώ. Ε, ε, ο Γκούνερ απευθύνθηκε σε μένα και θέλω να απαντήσω. Λες ότι υπάρχουν... Γκούνερ άκουσε με, σε σένα μιλάω. Ε, μίλησες για τις φτωχές χώρες. Δεν πιστεύω στο multitasking, ε, στην ταυτόχρονη επιτέλους διαφόρων ε, καθηκόντων. Ποιος μπορεί να πει τι θα γίνει με το φόρο, δηλαδή το 0,1%. Ποιο μπορεί να πει ότι θα είναι επιβλαβέ για το ε, κυρίαρχο ε, το, χρέο, το δημοσιονομικό χρέο δηλαδή των κρατών. Δηλαδή έχει μια διέστηση και εμεί πρέπει να βασιστούμε σε αυτό. Ε, ε Είπε ότι βοηθάνε οι βραχυπρόθεσμε σε χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Και πάλι εδώ είναι θεολογικού χαρακτήρα αυτή η δήλωση γιατί οι συναλλαγές υψηλή συχνότητας και οι βραχυπρόθυμες συναλλαγές αποσταθεροποιούν. Οπότε και πάλι εδώ γιατί να μην κάνουμε μια μελέτη πριν κάνουμε τέτοιους ισχυρισμούς. Ε, τρίτον και το πιο σημαντικό, ε, είπες ότι δεν θα μετακινηθούν οι άνθρωποι, οι συναλλαγές. Ωραία, ας φορολογήσουμε τους πολίτες. Για άντε να εντοπίσεις τους δικούς σου εκλογείς, ε, πόσο δίκαιο είναι αυτό, γιατί θα υπάρχουν ε, ε, καταχρήσεις όπως είπες, ε, αν πει σε παραδείγματο χάρη, ε, λε ότι επειδή δεν καταφέρνουμε να προσδιορίσουμε τη φορολογική βάση, θα πρέπει να απόσχουμε από την επιβολή οποιοδήποτε φόρου. Όχι, πρέπει να το αναλύσουμε και για τις ε, συναλλαγές ε, με ονομαστική αξία στα ευρώ, μα είναι εύκολο να τις εντοπίσουμε, ακόμη και αν γίνονται σε άλλες πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, μετά λες ότι αυτό δεν θα ε, παρεμποδίσει τις βραχυπρόθεσμες ή μεσοπρόθεσμες ε, ε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές γιατί θα είναι υψηλότερε από τον φόρο. Μάλιστα αυτό είναι καλό επιχείρημα υπέρ του φόρου γιατί θα έχουμε καλά έσοδα και δεν θα επιβαρύνουμε το φορολογικό σύστημα. Μα αποφάσισε με ποιον είσαι. Ε, εάν θέλουμε αυτό το φόρο, τι εννοείς, θα εκλείψουν οι συναλλαγές ή όχι. Αν παραμείνουν οι συναλλαγές στην Ευρώπη, γιατί να μην επιβάλλουμε το φόρο, δεν το καταλαβαίνω. Μην ξεχνάμε ότι ο, ο στόχος αυτού του φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα και ενδεχομένω να επηρεάσουμε και τον αριθμό των ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δεν συμφωνώ με αυτά που είπε για τον όγκο των συναλλαγών ότι είναι 10 φορέ υψηλότερο από την πραγματική οικονομία. Ε, αν μπορεί να επιχειρηματολογήσεις ε, και αν μπορεί να βασιστεί σε συγκεκριμένα στοιχεία, είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια σου. Άμα να μου πει ότι οι συναλλαγές είναι 10-15 φορέ υψηλότερε από την πραγματική οικονομία, αν μπορεί να μου προτάξει τέτοια επιχειρήματα τότε να κάνουμε μια καλή συζήτηση. Το πρόβλημα είναι ότι εσύ και άλλοι πετάτε μια δήλωση και δεν έχετε ε, προ υποστήριξή τη κανένα στοιχείο. Λοιπόν, τε, τελευταίο στοιχείο και αναφέρομαι και σε σένα και στη Βίκη. Λοιπόν, τι εννοεί ουσιαστικά ε, λέγοντας αυτά που λες. Ότι η διακυβέρνηση Ε, ότι οι διαχειριστές ε, πρέπει, ε, πρέπει να ελέγχουμε τους διαχειριστές γιατί δεν έχουν σωστή συμπεριφορά και πρέπει να έχουμε μία ομόσπονδη δομή όπως παραδείγματος χάρη η Επιτροπή των Σοφών που είχαμε παλιά για να ελέγξουν τους διαχειριστές. Ε, και οι αγορέ λέτε μάλιστα κάνουν και κάποια λάθη αλλά ε, γενικότερα συμπεριφέρονται καλά. Ε, ξέρετε, μην ξεχνάμε ότι οι αγορέ έχουν καταδείξει πρώτον ότι δεν έχουν καμία λογική και δεύτερον ότι οι βλάβες που προκαλούν είναι πελώριες γιατί δεν ε, ε, υποχρέωσαν οι κυβερνήσεις να επενδύσουμε στα, στα ενυπόθηκα δάνεια και δεν μας οδήγησαν αυτές ε, στην κρίση. Κανείς δεν ναι, τους υποχρέωσε να χρησιμοποιήσουν ε, αυτές τις υποδομές, τα παράγωγα κτλ. Γιατί δεν επενδύσανε στην πραγματική οικονομία. Ε, μπορεί να είναι πρόβλημα πολιτικής, αλλά οι αγορές αποφάσισαν να καταχραστούν των μέσων που είχαν στη διάθεσή τους. Και διαφωνώ, διαφωνώ μαζί Δεν λέω ότι είναι τέλειε οι κυβερνήσει, μα δεν είναι. Γιατί άνθρωποι κρύβονται πίσω από αυτά. Το θέμα είναι ότι οι κυβερνήσει ε, θα πρέπει να λογοδοτούν τελικά στους ε, ψηφοφόρου του ε, Και ποτέ όμω δεν λογοδοτούν οι αγορέ. Ποτέ. Sorry, sorry. we don't normally δεν μπορεί κάποιος να επανέλθει επί ζητήματος που είπε κάποιος άλλος να μου βάλει λόγια και μετά να κλείνει το θέμα. Θα την κλείσω τη συζήτηση, λέει ο, η Πρόεδρος, γιατί δεν νομίζω ότι είναι νόημο να έχουμε ε, παρεμβάσεις σαν εκρεμές από μερικούς. Όλοι επιχειρηματολογήσαμε υπέρ περισσότερων πληροφοριών, μελετών και ούτω καθεξής για να ληφθεί πολιτική απόφαση, όπως είπε και ο κύριος Γκοζές, γιατί εν τέλει λαμβάνονται πολιτικής υφής αποφάσεις. Ας μην μπούμε σε μια ιδεολογική συζήτηση. Εγώ δεν ήμουν ποτέ υπέρ ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Όμως η δική μου αντιπροσωπεία αποφάσισε ότι υπάρχει έσοδο από ένα τέτοιο φόρο, πέρα από τα μπόνους που δίνονται στα Golden Boys. Είτε πρόκειται για χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, δραστηριοτήτων και ούτω καθεξή. Θα ήθελα να πω, λέει ο κύριος Χέκμαρκ, ότι τα επιχειρήματά μου δεν ήταν ιδεολογικής υφής ήταν πραγματιστικής υφής. Το ζήτημα είναι κατά πόσο είναι λειτουργικό αυτό το πλαίσιο. Ναι, λέει η Πρόεδρος, αλλά όπως είπα κυρία Χακμάρκ, χρειαζόμαστε αποδεικτικά στοιχεία για να δούμε τι είναι εφικτό και τι όχι. Και θα ήθελα να ζητήσω από την κύρια Πόδηματά να μιλήσει επί ορισμένων συμπερασμάτων. Η κυρία Ποδηματά έχει το λόγο. Αν και συνόψισες πολύ καλά τη συζήτηση, θέλω να πω ότι παρά τις ε, διαφορετικές απόψεις, πραγματικά χαίρομαι το επίπεδο της συζήτησης που έγινε σε αυτή την Επιτροπή. Ε, ήταν εξαιρετικά υψηλό, εξαιρετικά χρήσιμο και νομίζω ότι ε, θα βοηθήσει πραγματικά την επίτευξη κάποιου συμβιβασμού. Άλλωστε, μέσω αυτής της Επιτροπής, αναφέρθηκε ο κύριος Γκοζές, στις ε, επιφυλάξεις που διατυπώνονταν όταν το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεση για τα, hedge funds. αντίστοιχε επιφυλάξεις το τελευταίο διάστημα έχουν ε, διατυπωθεί πολλές φορές για την ε, φιλόδοξη στάση που κρατάει το Κοινοβούλιο. Επιφυλάξεις υπήρχαν ισχυρές και όταν συζητάγαμε το πακέτο της χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Ε, εύχομαι και ελπίζω και σε αυτή την περίπτωση το Κοινοβούλιο, πέρα και ανεξάρτητα από ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις, διότι συμφωνώ και εγώ ε, ότι το ζήτημα δεν είναι ε, ιδεολογικό. Το ζήτημα είναι ζήτημα ευρωπαϊκό πρωτίστως κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό και ανέφερα πριν ότι είμαστε σε μια ιδιαίτερη συγκυρία μιας πρωτοφανούς κρίσης. Συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει ανάγκη αναζήτησης ε, νέων πόρων, νέων πόρων για την κοινότητα, νέων πόρων για τους εθνικούς προϋπολογισμούς και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε επίσης ότι το κύριο βάρος δεν μπορεί να, όχι το κύριο, το αποκλειστικό βάρος δεν μπορεί να συνεχίσει ε, να βρίσκεται στους ώμους των καταναλωτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Άρα το ζήτημα δεν είναι ένας ακόμα φόρος, το ζήτημα είναι ε, ένας δικαιότερος καταμερισμός των φορολογικών βαρών και η φορολόγηση ε, ενός τομέα που έως σήμερα εξαιρείται κατά βάση, κατά τεκμήριο από τη φορολόγηση, όπως είναι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, και σε αυτό το πλαίσιο της ανάγκης να ενταχθεί στις υποχρεώσεις φορολόγησης και ο τομέας αυτός, λέω ότι η καλύτερη δυνατή επιλογή στη σημερινή συγκυρία είναι η επιλογή ενός φόρου που θα μπορεί να επηρεάζει και τις συμπεριφορές, να αποθαλύνει τις μολυντικές, τις επιβαρυντικές συμπεριφορές. Γι' αυτό συζητάμε ασχέτως της ιδιαίτερης οπτικής μας γωνίας, οπτικής μας και για την φορολόγηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, τη φορολόγηση του τη φορολόγηση του ενεργειακού μείγματος. Ε, αναζητούμε ε, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, νέους φόρους που θα μπορούν να επηρεάσουν, να αποτρέπουν, να αποθαρρύνουν επιβλαβείς συμπεριφορές. Ε, και σε τελευταία ανάλυση μεταξύ της επιλογής της φορολόγησης του κέρδους που είναι η συζήτηση όλη που γίνεται για την ε, φορολόγηση του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι μεταξύ αυτής της επιλογής ε, και της επιλογής φορολόγησης και άρα αποθάρρυνση της κερδοσκοπίας είναι προτιμότερο να εστιάσουμε την προσοχή μας στην φορολόγηση της κερδοσκοπίας παρά στη φορολόγηση του φόρους και του, ε, του κέρδους. Και, εν πάση περιπτώσει, ε, στις παρατηρήσεις και στις ανησυχίες ορισμένων συναδέλφων ότι θα πλήξει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θα διώξει τις συναλλαγές ε, εκτός Ευρώπης. Ένα επιχείρημα ε, ακούστηκε πριν ότι ε, δεν μπορεί να μην συνυπολογίζουμε καθόλου το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούν να φύγουν οι πολίτες που υφίστανται σήμερα τα φορολογικά βάρη παντού στην Ευρώπη, στη χώρα μου και αλλού, ε, φεύγουν επενδύσεις σε μια εποχή ιδιαίτερα δύσκολη, πρωτοφανούς ύφεση, διότι ο φόρος επί των επιχειρήσεων είναι εξαιρετικά υψηλός και είναι εξαιρετικά υψηλός λόγω αυτής της τιστάνιας προσπάθειας αύξησης των εσόδων, ούτω ώστε να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αλλά δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Στην Ελλάδα γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για την αύξηση του, φόρου, ε, του επιχειρηματικού φόρου πάνω από το 12,5%. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο εκεί. Ξαναλέω, πέρα από ιδεολογικοπολιτικές τοποθετήσεις, έχουμε υποχρέωση, κατά τη γνώμη μου, να στραφούμε σε άλλες κατευθύνσεις, προκειμένου να δώσουμε στους πολίτες ένα μήνυμα ότι αυτό το Κοινοβούλιο θέλει και μπορεί να αναζητήσει εναλλακτικέ συνυπολογίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ όλους για τις παρατηρήσεις σας. Ε, δεν είχατε, φαντάζομαι, περισσότερο τον χρόνο να δείτε τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Φαντάζομαι ότι θα το κάνετε και θα ε, προχωρήσουμε σε μια νέα συνάντηση των σκιωδών ε, στην, στη διάρκεια της επόμενης Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ πολύ, Αλή. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε στις 25 Ιανουαρίου στην Επιτροπή, άρα έχετε χρόνο να συνομιλήσετε με τους σκιώδης για ενδεχόμενους συμβασμούς και στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι για την υπομονή σας, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Έχουμε δύο τώρα γνωμοδοτήσεις, στο μέλλον των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Η κυρία Οκονή είναι παρούσα και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις, διότι συνεισέφεραν σε αυτή την εργασία η Επιτροπή ΕΚΟΝ εργάζεται επί μίας γνωμοδότησης για μία έκθεση όπου η Επιτροπή Απασχόλησης είναι αρμόδια επί της ουσίας. Εργαστήκαμε επί όλων των συστημάτων που σχετίζονται με τις κρατικές επιδοτήσεις. Καταρχήν θα ήθελα να πω σε σχέση με το σύνολο των συζητήσεων που έλαβαν χώρα εδώ στο Κοινοβούλιο, δηλαδή τις ανταλλαγές απόψεων στις Ολομέλειες ή ως προς το Φόρουμ για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Ενδιαφέροντος που οργάνωσε η, Βελγική Προεδρία, θα ήθελα να πω ότι απορρέει μια πολιτική διάσταση αυτής της συλλογιστικής για τις δημόσιες υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια της κρίσης. Θα ήθελα να πω ότι αυτές οι κοινωνικές ε, υπηρεσίες βοήθησαν για την υπερπίδηση της κρίσης και εκπροσωπούν το 9,5% της συνολικής απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα επιβεβαιώνουν μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. τα κείμενα επί των οποίων βασιστήκαμε δεν έχουν την επαρκή νομική διαφάνεια και γι' αυτό θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τα κείμενα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη απέστειλε ένα μήνυμα με το Single Market Act όπου οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να ενταχθούν σε μία ανακοίνωση γενικότερου ενδιαφέροντος που αναμένουμε με αδημονία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν νομική ε, διαφάνεια, γι' αυτό προβήκαμε σε προσαρμογές. Πολλές φορές εφαρμόζουμε στις κοινωνικές υπηρεσίες κανόνες που ισχύουν για οι οικονομικές υπηρεσίες που δεν εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Για να διασαφηνίσουμε το όλο πλαίσιο, αρχίζουμε με μία πτυχή του θέματος που είναι ύψης της ε, σημασίας. Εγώ μιλώ για μία μεθοδολογία και βλέπω ότι στην πράξη ενιαίας αγοράς η Επιτροπή μιλάει για μία εργαλειοθήκη. Άρα συμμεριζόμαστε αυτή την σκέψη μέσα στα πλαίσια μίας ανακοίνωσης που αναμένουμε. Χαίρομαι για αυτές τις εξελίξεις κατά συνέπεια σε σχέση με το σημείο τρία αυτής της και επειδή πρόκειται για ελάχιστους κανόνες, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να μελετήσουμε μία ελάχιστη διευθέτηση, διότι σήμερα δεν υφίσταται και θα πρέπει να ορίσουμε ένα ποσοτικό κατόφλι θα πρέπει λοιπόν να απλουστεύσουμε τις διαδικασίες στους παρόχους υπηρεσιών και να επιτρέψουμε στις επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ να μπορέσουν να παρέμβουν για αυτού του τύπου διαδικασίες. Τέταρτον, ως προς τη διαδικασία κοινοποίησης στα πλαίσια της διαδικασίας ε, επικύρωσης για τους ε, πάροχους υπηρεσιών, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τονίσει ότι απαλλάσσονται της κοινοποιήσεως ορισμένοι παρεμβαίνονται στην αγορά. Θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει την ε, έννοια των οικονομικών συναλλαγών σε σχέση με κείμενα τα οποία δεν είναι σαφή επ' αυτού. Το πακέτο Monty Cruz δεν αφορούν παρά οικονομικές δραστηριότητες, άρα οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν εντάσσονται εδώ. Δεν βρίσκουν τη σωστή τους θέση εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τα κείμενα που την χάνουν εφαρμογή σε αυτόν τον τομέα. Για το σημείο 6 θα θέλαμε να αντιστραφεί ο φόρτος σε σχέση με την υπέραντη στάθμιση στα πλαίσια αυτής της απλούστευσης διαδικασιών θα κρίνουμε σκόπιμο να αντιστραφεί αυτό το άχθος και ο έλεγχος της υπεραντιστάθμισης να σχετίζεται με μία ε, πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση του παρόχου. Σήμερα οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι βιώσιμες παρά μόνον εάν αρθεί αυτή η νομική αβεβαιότητα και διασαφηνίσουμε κάπως τα κείμενα. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται το, το κείμενο μαζί με την Επιτροπή ε, Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ο Πίτερ Σάιμον θα λάβει ο, το λόγο και μετά η Σοφή Ιντβέλτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε όλοι πλήρη συνέστηση του θέματος. Οι υπηρεσίες ε, για τις οποίες συζητούμε είναι, επηρεάζουν την καθημερινότητα του καθενός μας, έχουν τεράστια σημασία, είτε πρόκειται για ε, φροντίδα παιδιών, είτε πρόκειται για ε, φροντίδα ηλικιωμένων κτλ. Η, χωρίς ε, αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες η κοινωνία μας θα ήταν φτωχότερη. Γι' αυτό πρέπει να προστατευθούν αυτές οι υπηρεσίες. Θα πρέπει να φτιάξουμε λοιπόν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο να τις προστατεύει και να τις, ε, να τις κάνει απλούστερες από ό,τι στο παρελθόν. Γιατί μέχρι σήμερα υπήρχε μια, ένα τεράστιο μπέρδεμα μεταξύ και των παρόχων αυτών των υπηρεσιών και όλων των άλλων ευδιο ενδιαφερομένων που το είδαμε σε κάποιες μελέτες και έρευνες που κάναμε στο παρελθόν. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Και εδώ βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς θα καταλήξουμε σε αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το γεγονός ότι έφτιαξε την εκθεσή της που είναι καλή βάση για συζήτηση αλλά θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα ε, αρκετά σημαντικά. Πρώτον, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι για τον, για τον ορισμό, τον οργάνωση και τη χρηματοδότηση ε, εδώ ε, υπάρχει εθνική αρμοδιότητα. αρχή της επικουρικότητας άρα πως το ξεπεράσουμε το θέμα αυτό από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε οι υπάροχοι υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες μοναχά στο τοπικό επίπεδο και ειδικά για τον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών υπάρχουν πάρα πολλές μικρομεσαίες ε, και μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αυτή τη δουλειά αυτοί οι υπάροχοι πρέπει να απαλλαχθούν, να εξαιρεθούν Επίσης πρέπει να συζητήσουμε το θέμα αντεμήνυμης που ανέφερε και η συγκεκριά να έχουμε μια ειδική ε, ρύθμιση εδώ να ορίσουμε αν θέλετε κατόφλια τεμήνυμης για τις κοινωνικές υπηρεσίες κάτι να κάνουμε τρίτο θέμα ε, το να αναφερθώ στις κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελία και θα ήθελα να τονίσω αυτό το κοινή ωφελία γενικού ενδιαφέροντος γιατί εδώ αυτό δημιουργεί και η διάκριση βέβαια αυτών των υπηρεσιών από τις υπηρεσίες α, τις οικονομικές αν θέλετε είναι πολύ σημαντικό να ε, συζητηθεί και να αποφασιστεί νομίζω ότι είναι κλείνοντα να πω ότι είναι πολύ καλή έκθεση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε μεγάλη συζήτηση και βοηθάει καλή συνεργασία στο μέλλον η Σόφιντ Φέλτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω κάποιες αμφιβολίες, όχι για την έκθεση αυτή καθεαυτή, αλλά για τη συζήτηση και την τροπή που παίρνει. Γιατί τη συζήτηση αυτή την έχουμε κάνει επανειλημμένα. Και το επιχείρημα, ας πούμε, που ακούσαμε, δημιου... Ε, ε, μας δημιουργεί πρόβλημα. Η συνθήκη λέει ότι οι εθνικές αρχές αποφασίζουν για την οργάνωση και τη χρηματοδότηση των ε, υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος. Όταν αρχίσουμε λοιπόν μια συζήτηση σαν και αυτή που φαίνεται να ξεκίνησε εδώ και αρχίζουμε και λέμε ότι κάποιοι πάροχοι υπηρεσιών, κάποιες υπηρεσίες πρέπει να εξαιρεθούν, τότε τι κάνουμε, μπαίνουμε στα χωράφια των εθνικών αρμοδιοτήτων. Ε, θίγεται η αρχή της επικουρικότητας που είναι το πρόβλημα το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν οριστεί ποτέ οι υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος και υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος κτλ. Αναφέρεται η φροντίδα των ηλικιωμένων. Μπορεί στη χώρα σας οι φροντίδες αυτές να παρέχονται αποκλειστικά από το δημόσιο. Σε άλλες χώρες όμως υπάρχει απελευθέρωση και εμπλέκεται και ο ιδιωτικό τομέα. Άμα θέλετε λοιπόν ε, να προχωρήσουμε θα πρέπει να δουθούν κάποιοι ορισμοί. Αλλά τη στιγμή που αρχίσουμε να δίνουμε ορισμούς για το ποιες υπηρεσίε είναι ποιες, αρχίζουμε και μπαίνουμε στο χωράφι και τις αρμοδιότητες των κρατών μελών επαναλαμβάνω αυτό που έχω πει επανειλημμένα πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες εφαρμογής της συνθήκης και για να τις διευκρινίσουμε πρέπει να ορίσουμε το πρόβλημα διότι γενικώ λέμε ότι οι κανόνες ε, της διατάξης της συνθήκης ε, ουσιαστικά ε, είναι τροχοπέδι για την εφαρμογή κοινωνικών και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά ξέρουμε και όλα πολύ καλά ότι είναι πιο εύκολο η παροχή υπηρεσιών να κάποιων υπηρεσιών τέλο πάντων να πάρουν εξαίρεση ε, από τους κανόνες της κρατικής ενίσχυσης κτλ. Μόλις βάλουμε το κοινωνικό, social, αμέσως υποτίθεται ότι βγαίνουμε από τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Χτες κουβεντιάζαμε την υπόθεση Google. Θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι οι μηχανές αναζήτησης είναι κοινωνικές υπηρεσίες. Διότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβηση στις α, ε, μηχανές αναζήτησης. Αλλά αυτές οι μηχανές αναζήτησης που μπορεί να είναι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να εξαιρούνται. Συγγνώμη. Καταλαβαίνετε τι εννοώ ότι αυτό θα πρέπει να δούμε πώς παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές με εμπορικό τρόπο, με οικονομικό τρόπο της αγοράς κτλ. Τέλος πάντων χρόνια ολόκληρα δουλεύω για το θέμα αυτό, ο σωστό ορισμό και σαφή ορισμό δεν βρήκα ακόμη, δεν είδα να προτείνεται και φοβάμαι ότι για πολλά χρόνια θα τα... Ε, θα αγωνιζόμαστε με αυτό. Ε, να του δώσω εγώ λίγο χρόνο στον συνάδελφο που ήθελε να μιλήσει. Όχι, λοιπόν. Ενδιαφέρουσα συζήτηση, δεν την κάνουμε πρώτη φορά, αλλά οι κριτικέ που κάνουμε θα πρέπει να είναι λίγο πιο συγκεκριμένε, γιατί εν προκειμένου κανεί δεν λέει ότι δεν θα χρειαζόταν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για να προσδιορίσουμε τους εφαρμοστέους κανόνες και ταυτόχρονα όμως να αφήσουμε μια ευελιξία, ένα περιθώριο ελιγμών στα κράτη-μέλη για να προσδιορίσουν την εμβέλεια των εξαιρέσεων. Κάθε κράτος δηλαδή θα προσδιορίσει το εύρος ε, των ε, εξαιρέσεων, αλλά αυτή τη στιγμή αποφασίσουμε ότι δεν ε, εφαρμόζεται εξαίρεση, όλοι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους, για τη χρηματοδότηση δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναθεωρήσει τους χρηματοδοτικούς κανόνες αλλά μιλάμε για χρηματοδότηση που δεν είναι κρατική επιδότηση. Οι προτάσεις ε, της ε, Σοφή ε, ακολουθούν τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, ζητάμε μεταξύ άλλων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τι επιπτώσει επί του ενδοκινοτικού εμπορίου. Τι ε, λέμε ουσιαστικά, ότι μία οντότητα ε, που θα δώσει χρηματοδότηση 70 εκατομμύρια το χρόνο για ένα κέντρο υποδοχή κακοποιημένων γυναικών θα επηρεάσει το ενδοκινοτικό εμπορίο και άρα πρέπει να υπαχθεί σε διάφορα κριτήρια για να αιτιολογήσουμε ότι δεν πρόκειται για κρατική Ευρωπαϊκή ε, επιδότηση. Αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να ε, ξεκινήσει ε, με μία ανάλυση για τις τράπεζες παρά την υψηλή χρηματοδότηση. Και δηλαδή μία τοπική αυτοδιοίκηση που θα δώσει 70 εκατομμύρια για το κέντρο υποδοχής κακοποιημένων γυναικών θα πούμε ότι στρεβλώνεται το ενδοκινοτικό εμπόριο λόγω αυτού. Μα συγγνώμη, είναι όλα ανάποδα. Πρέπει να δούμε τι είναι διασυνοριακό, τι είναι κοινή ωφελία, τι είναι τοπικού, τοπικής ωφελία, ποια υπηρεσία είναι τοπική ωφελία. Αυτό το κέντρο υποδοχή ε, που λαμβάνει την επιδότηση ε, στην Ολλανδία ή στη Γαλλία από ε, μια τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ανταγωνισμό. δεν τίθεται θέμα ευρωπαϊκής αγοράς. Για τα διασυνοριακά μιλάμε. Αναρωτιόμαστε αν ε, θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με αυτό. Μήπω ε, επιφέρουμε ένα επιπρόσθετο άχρηστο όμω γραφειοκρατικό άχθο αντί να ε, βελτιώσουμε την κατάσταση. Οι προτάσει που βλέπουμε μέσα στην έκθεση πάντω είναι σωστέ. Και στην Επιτροπή της Εσωτερικής Αγοράς την ίδια στάση θα κρατήσω εγώ θα υπερασπιστώ αυτές και παρεμφερείς προτάσεις. Σήμερα έχουμε ένα ε, χρονοδιάγραμμα που όλο ένα και συγκεκριμενοποιείται. Ε, ο πρόεδρος Μπαρόζο ε, στην εκστρατεία του για, να, για την Προεδρία το είχε ανακοινώσει αυτό ότι είναι πήγον, πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κάποιοι σοσιαλιστές συνάδελφοι είπαν μάλιστα αφού το λέει εντάξει θα το κάνουμε. Θα ε, εντάξει, ε, πρέπει να πολιτικοποιήσω το θέμα γιατί εκνευρίζομαι. Ε, είπαμε το 2011 θα γίνει. Ωραία. Μόλις βγήκε το σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2010, ξαφνικά μεταφέρθηκαν τα μέτρα για το 2011. Αλλά τώρα όμως το πρόγραμμα του 2011 δεν υπάρχει τίποτα και αναβάλλεται για το 2012. Ε, μα, ε, συγγνώμη, δεν τηρούμε ε, τις υποσχέσεις μας, δεν είναι λογικό. Ε, άλλα υποσχέθηκε ο κύριος Μπαρόσο και πρέπει να τα καταγγείλουμε αυτά χρησιμοποιώντα αυτό το συγκεκριμένο θέμα για τις υπηρεσίες ε, κοινή ε, ωφελίας, ο κύριος ε, Γκοζάς. Ε, συντομία για να συγχαρώ ε, ε, τον εισηγητή για την έκθεση, ε, την εισηγήτρια για την έκθεση. Συμφωνώ με τη Σοφή όταν λέει ότι δύσκολα μπορούμε να προσδιορίσουμε τα κριτήρια, αλλά συμφωνώ και με τον Πασκάλ. Ε, λέει ότι είναι θέμα κρατικό, θέμα τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να έχουμε κάποια συνέπεια. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα ανάλογα με τη χώρα και πολλέ υπηρεσίε, κοινωνικέ υπηρεσίε, δηλαδή που βοηθούν τους ανθρώπους ε, ε, χρηματοδοτούνται από τις δημόσιες δαπάνες, από τις κρατικές επιδοτήσεις, πολλές από αυτές. Οπότε ε, δεν θα πρέπει να παρισφρεί σε αυτό το τομέα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό γιατί είναι κακό για την εικόνα της Ευρώπης. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε το σπίτι σας γιατί μας εμποδίζει η Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ξέρετε ότι είμαι φιλοευρωπαϊστής. Υπάρχουν τομείς όπου πρέπει να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εδώ πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι ε, ούτω ώστε να μην ανατρέψουμε την ε, κατάσταση που υπάρχει στα κράτη-μέλη. Δεν χρηματοδοτούν όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο τι κοινωνικέ υπηρεσίε και δεν έχουν τα ίδια αποτελέσματα. Αντιπαραβάλλεται την κατάσταση ε, στη Γαλλία και στο Βέλγιο, γειτονικέ χώρε. Υπάρχει μια φήμη στη Γαλλία που λέει ότι ε, υπάρχει καλύτερη περίθαλψη, είναι πιο φτηνή στο Βέλγιο, έτσι, σε σχέση με τη Γαλλία. Ωραία. Ε, πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά σε αυτό το τομέα δεν πρέπει με συστηματικό τρόπο να παρεμβαίνουμε. Ε, μην ξεχνάτε την επικουρικότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας δώσω το λόγο. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω όμως ότι δεν έχουμε χρόνο και έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την επικουρικότητα. Δίνω μεγάλη μάχη για την επικουρικότητα. Διότι μιλάμε για μία εξισορρόπηση και νομίζω ότι οι αρμοδιότητες πιέζουν ε, ως προς την επικουρικότητα. με βάση το πακέτο Monty Cruz βλέπουμε ότι αυτές οι ενδείξεις δεν αρκούν. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι ίσως την επόμενη μέρα η Κομισιόν κάνει προσφυγή στο ΔΕΚ τάχει γιατί πρέπει να φύγω κι εγώ. Θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές το εξή. Όταν ήταν εδώ κύριε, κύριε Γκοζές, όταν ήμασταν εδώ χρόνια πριν, είχαμε αποφασίσει ότι αποκλείονται ορισμένες υπηρεσίες από τη διαδικασία κοινοποίησης. Δηλαδή όταν υπάρχουν 100 εκατομμύρια τζίρος, τότε αποκλείονται αυτοί οι πάροχοι. Άρα δεν μιλάμε για θύματα ε, η, βίας. Μιλάμε για νοσοκομεία τα οποία είναι κερδοφόρα. Μιλάμε για κοινωνική στέγη, όπως ισχύει στη χώρα μου, το που αποτελεί κοινωνική υπηρεσία και οι πάροχοι έχουν κατά 60% εμπορικές δραστηριότητες, αλλά έχουν κρατικές, δέχονται κρατικές ενισχύσεις, διότι η συνθήκη ακριβώς αυτό αναφέρει ότι θα πρέπει να δούμε τον αθέμητο διασυνοριακό ανταγωνισμό. Αλλά όλα αυτά έχουν διασαφινιστεί. Εάν ισχύσουν δικοί κανόνες για τις κοινωνικές υπηρεσίες ε, κοινωνικού, γενικού ενδιαφέροντος είναι θα πρέπει να τις οριοθετήσουμε, αλλά οργανώνονται διαφορετικά στις διαφορετικές χώρες. Αν πούμε ότι για αυτή την, ε, τον κατάλογο θα πρέπει να υπάρχει κοινωνική στέγαση, αυτό σημαίνει ότι η χώρα μου θα πρέπει να ε, οργανώσει εκ νέου την κοινωνική στέγη, διότι κατά 60% οργανώνεται από τον εμπορικό τομέα. Κύριε ε, Ρονκόνη, θα ο θα έχετε μεγάλες δυσκολίες με τους σκιώδεις. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Θα ήθελα πω στη Σοφή ότι γνωρίζω τη διαδικασία αυτού του θέματος και ξέρω ότι η δική σας πολιτική είναι διαφορετική και δεν μπορείτε να προβείτε σε κατεξουδότηση πράξη σε άλλους φορείς. Αλλά δεν πρέπει να κάνουμε και τίποτα. Εμείς λέμε ότι στις δικές μας περιφέρειες υπάρχει ε, διαφορετική διαχείριση του θέματος. Θα πρέπει λοιπόν να διασαφηνίσουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους υπάρχοντες κανόνες, να δούμε πού μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδομητικά. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 15 Δεκεμβρίου, τα υπόλοιπα 7 λεπτά θα δούμε τη γνωμοδότηση που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας υπηρεσιών και θα πρέπει να υποβληθεί αυτή η γνωμοδότηση στα αγγλικά καθώς και οι τροπολογίες μέχρι τις 7 ε, Δεκεμβρίου, διότι ε, έχουμε μείνει πολύ πίσω. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντω ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο για αυτό το κείμενο για τη μεταφορά της οδηγίας. Δεν έχουμε χρόνο γιατί η ΙΜΚΟ είναι καθήλυνα αρμόδια και θα εγκρίνει την έκθεση τον Ιανουάριο 2011 και άρα έπρεπε να ε, γνωμοδοτήσει η ΕΚΟΝ ε, πολύ νωρίτερα. Ε, ζητώ συγγνώμη για το στενό χρονοδιάγραμμα. Με ρωτήσατε τώρα γιατί. Ε, σας είπα, η ΙΜΚΟ είναι η επί της αρμόδια επιτροπή και ο τομέας αυτών των υπηρεσιών ε, έχει μέγιστη σημασία για την οικονομία, για την καταπολέμηση της ε, ανεργίας, 70% του ΑΕΠ, ε, 15% των θέσεων απασχόλησης, 40% ε, ε, του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και 40% των θέσεων απασχόλησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις ε, υπηρεσίες, άρα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Το 2006 εργάστηκε πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 2011 είναι σημαντικό να ακολουθήσει την, να παρακολουθήσει τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στην Εθνική νομοθεσία. Εκεί ε, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι ε, προσδοκούσαμε. Και αυτό λέω μέσα στη γνωμοδότηση ότι πρέπει να υπολογίσουμε και την περιπλοκότητα της μεταφοράς της οδηγίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα στη Γαλλία. Η μεταφορά στην γαλλική νομοθεσία ε, δεν γίνεται βάση ενιαίου εγγραφού. Υπάρχουν πολλά και διαφορετικά για κάθε ένα επιμέρου σημείο της εφαρμογής. Ε, γι' αυτό ε, και είναι μακροσκελής εργασία και γι' αυτό είναι περίπλοκη. Και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και σε άλλα κράτη-μέλη. Οπότε, για να διαφυλάξουμε την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών ε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε βέλτιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες ε, και ε, μέσω της, των μονοαπευθυντικών θηρίδων να αυξήσουμε και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε στην ηλεκτρονική οδό, θα ήταν ενδεδειγμένο να χορηγήσουμε για τους παρόχους πρόσβασης υπηρεσίες άλλων κρατών μέσω μιας απλούστευσης της προσβασιμότητας. Τι εννοώ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβεβαιώσουμε ότι αυτές οι μονοαπευθυντικές ε, θηρίδες είναι το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο, ούτως ώστε οι μικρές επιχειρήσεις και οι μεγάλες εξάλλου, ε, να μπορέσουν να παράσχουν υπηρεσίες στην επικράτεια άλλων κρατών. Αυτή η μονοαπευθυντική θερίδα λοιπόν έτσι φαίνεται να είναι το πλέον ενδεδειγμένο εργαλείο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Να διευκρινίσουμε επίση το πεδίο εφαρμογή. Το άρθρο 2 τη οδηγία αποκλεί τι τις μη οικονομικέ υπηρεσίε. Είναι δύσκολο να ριοθετήσουμε τις υπηρεσίες και ζητούμε εδώ ακριβώς αυτό, τη διευκρίνηση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Λοιπόν, για τη μεταφορά τώρα, Εξυπακούτε ότι πρέπει να προχωρήσουμε, να προβούμε στην εφαρμογή. Ε, αλλά υπάρχει αμοιβαία αξιολόγηση που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Δηλαδή, Χρειάζεται ανάλυση από κάθε κράτος μέλος και από την Επιτροπή και να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης ούτω ώστε να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο για την πρόοδο που σημειώνεται για τη μεταφορά της οδηγίας και για την ποιότητα της μεταφοράς ε, στις εθνικές νομοθεσίες. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκπονήσει μία έκθεση για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Κατακλείδη. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με την ε, εφαρμογή και είναι σημαντικό να τοποθετηθεί και το Κοινοβούλιο. Γιατί, διότι λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η μεταφορά αυτής της οδηγίας στην Ευρώπη θα ε, εκπροσωπούσε σε 1,5% το ΑΕΠ επιπρόσθετο έτσι σε σχέση θα δημιουργούσε άλλο 1,5% ε, του ΑΕΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν εφαρμοζόταν σωστά. Γι' αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό το Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να ενημερώνεται και να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, τη μεταφορά της οδηγίας και κυρίως την ποιότητα της μεταφοράς. Ο κύριος και ο Διέχουμε μόνο που έχει ζητήσει το λόγο. Θέλετε το Και εγώ παρακολουθώ αυτό το θέμα από πλευράς Επιτροπής. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι υπάρχει συνένεση σε επίπεδο ΙΜΚΟ διότι σε αντίθεση με αυτά που λέει η Κομισιόν με βάση το Single Market Act, και αυτό το ξέρει η κυρία Οκονή, είναι ότι ο Μισελ Μπαρνιέ μιλά για δύο ή τρία, τρεις μονάδες ε, αναπτυξιακής πορείας. Το ζήτημα είναι όμως να δούμε τι προστιθέμενη αξία μας ε, δίνει η υπηρεσία αυτή με βάση το ΑΕΠ. Νομίζω ότι είναι πρόωρο να αποτιμήσουμε το, τον αντίκτυπο της, υπηρεσίας, της οδηγίας περί υπηρεσιών, γιατί υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις και αν δούμε τις ε, πρώτες εκτιμήσεις, βλέπουμε ότι αυτό που μετρά δεν είναι το μακροοικονομικό πλαίσιο, αλλά η εφαρμογή της οδηγίας περί υπηρεσιών. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτεροι ε, προσεκτικοί σε σχέση με το ΑΕΠ και τον δίκτυ απασχόλησης σε αυτή την εκτίμηση και με βάση ιδιαίτερα το Single Market Act. Σε σχέση με τη συζήτηση στην ΙΜΚΟ, θα πρέπει να δούμε τι πληροφορίες διαθέτουμε και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο υπάρχουν επιχειρήσεις που θέλουν να προωθήσουν μία δραστηριότητα σε άλλες χώρες. Αυτό το βλέπουμε και μέσα στα πλαίσια της ΕΚΟΝ. Θα πρέπει ίσως να ε, ε, διευρύνουμε την μονοαπευθυντική θηρίδα και θα πρέπει να ασχοληθούμε και με θέματα εργατικού δικαίου, διότι ένα από τα θέματα που μας απασχόλησε αφορούσε τη χώρα προέλευσης. Και αυτό που μας ενδιέφερε ήταν ε, η αρχική έκδοση της οδηγίας και τα πλαίσια αυτά δεν αφορούν κανόνες ε, πρόσβασης στην αγορά σε σχέση με την ασφάλεια τύπου προϊόντος και λοιπά, αλλά μιλάμε για μια διαδικασία αδειοδότησης με βάση το φορολογικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι τι πληροφορίες διατίθενται στους ε, παρόχους για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε αυτά τα επιμέρους ε, ζητήματα. Αυτές είναι οι δύο βασικές παρατηρήσεις που θα ήθελα να κάνω έτσι ώστε να φτάσουμε σε έναν εύλογο συμβιβασμό θέλετε να επανέλθετε διότι έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Μπορείτε να μιλήσετε αργότερα ίσως. Οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν στα αγγλικά μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου και μετά θα ψηφίσουμε στις 13. Και αυτή είναι και η τελική πληροφορία. Σύ στις 13 Δεκεμβρίου την Δευτέρα σας. Θα συνεδριάσουμε σε 7 το βράδυ. Σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.